Uh, um, Γεια σας. Θα κηρύξω επίσημα την έναρξη ε, των εργασιών γιατί με ειδοποιούν ότι ο κύριος Μάγερ, που είναι η πρώτη έκθεση έχει φύγει από το γραφείο του οπότε μέχρι να φτάσει θα σας πω τα πρώτα και τα διαδικαστικά. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου. Ε, είναι σήμερα το απόγευμα και αύριο ε, δύο πλήρης συνεδριάσεις και έχουμε και ψηφοφορία στις 10 παρατέταρτο με κάποιες αποφάσεις για επίσημα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου για το νέο νομοθετικό πλαίσιο, όλη αυτή τη δέσμη, καθώς επίσης και για εντολή που θα πρέπει να ψηφίσουμε για διάφορα θέματα ασφάλειας των καταναλωτών και προϊόντων να είστε στην ώρα σας. Όπως πάντα μεταδίδεται η συνεδρίαση μας στο διαδίκτυο και καλωσορίζω όλους τους τηλεθεατές στο webcast. Και νομίζω ότι έχουμε και νέο newsletter αν δεν απατώμε. Α, όχι ακόμα. Ε, προσεχώς τότε. Ε, όχι ακόμα. Αν θέλετε το παλιό, ε, του περασμένου μήνα είναι στην ιστοσελίδα. Επίσης θέλω να σας πω ότι αύριο το απόγευμα στις 3.30 παρένθεση σας θυμίζω ότι αύριο το απόγευμα ε, θα ακούσουμε ε, στη διάσκεψη των Προέδρων τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα αρχίσουμε ε, την απογευματινή συνεδρίαση όχι στις 3 αλλά στις 3.30 και θα τελειώσουμε 6 παρατέταρτο και ακολουθούν συντονιστές μέχρι τις 9 τις 19, συγγνώμη, τις 7. Λοιπόν, αύριο στις 3.30 θα γίνει σημαντική ακρόαση και θα ε, προεδρεύσει και ο κύριος ε, Μάγερ, είναι τα θέματα των επιβατών, των ταξιδιών και η πρόταση ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Επιτροπή μας. Ένα τελευταίο, πριν εγκρίνουμε επισήμω και την ημερήσια διάταξη, είναι το εξή. Περιμένουμε τη γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής για την αναδιατύπωση ε, της πρόταση για εναρμόνιση των μηχανημάτων υποπίεση δεν είναι στη σημερινή ημερήσια διάταξη παρόλο που ήταν αναμενόμενο. Λοιπόν, συμφωνείτε με το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης όπως έχει προταθεί. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Μερικές ε, ακόμα ενημερωτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, για το πρόγραμμα καταναλωτών 2014-2020 βλέπω εδώ παρόντα τον εισηγητή μας τον κύριο Ροσφόρ. Αντί να κάνω εγώ την ανακοίνωση, θέλετε εσείς μήπως να συνοψίσετε τη συμφωνία μας για το πρόγραμμα που θα υποβάλουμε αύριο στην Επιτροπή. Ah, ναι, κύριε Πρόεδρε. Όλα καλά πήγαν. Αυτός ο τριμερής ε, διάλογος ε, επέτρεψε ένα θετικό αποτέλεσμα. Καταφέραμε να καταλήξουμε συμβιβασμό όσον αφορά τις ε, κατεξιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις. Ήσασταν ε, ένας από τους βασικούς ε, παίκτες ε, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, γιατί κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα κάνουμε και κάποιο είδους απολογισμό και τότε θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι οι βασικές διατάξεις θα έχουν όντως σωστά εφαρμοστεί ή θα ενημερωθούμε για τα προγράμματα τα οποία ε, δεν ε, έχουν εφαρμοστεί αυτά τα δύο πρώτα χρόνια. Θα έχουμε λοιπόν ε, επικές συζητήσεις, έξι μήνες, οκτώ μήνες, ένα χρόνο για να καταλήξουμε τελικά ότι θα πρέπει η τρίτη χρονιά, ε, που είναι η βασική χρονιά, να μας δίνει τη δυνατότητα αξιολόγηση της πρώτης χρονιάς, ε, για να μπορέσουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς ε, να ολοκληρώσουμε τις τροποποιήσεις για τα προγράμματα των δύο ετών που, μένουν ακόμη να εφαρμοστούν. Ελπίζω ότι όλα αυτά θα εκτιμηθούν δεόντως από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ε, πολύ καλή σας ε, παρουσίαση των ε, συμβιβασμών. Αύριο θα το εγκρίνουμε αυτό. Ελπίζω ότι θα είναι θετική η ψηφοφορία αύριο. Δύο ακόμα ενημερωτικά. Πρώτον, να σας ενημερώσω ότι είμαστε μία πιλωτική επιτροπή για τις συνεδριάσεις χωρίς ε, έγγραφα χωρίς ε, ε, χαρτιά. Αν το δείτε, αν δείτε και το νηστό τοπό μας, θα καταλάβετε ότι μπορείτε εκεί να λάβετε όλα τα στοιχεία, όλα τα έγγραφα των ε, συνεδριάσεών μας ε, αντί να έχετε την τεράστια χαρτούρα που βλέπετε τώρα μπροστά σας, το φάκελό σας. Ελπίζουμε να πάει καλά αυτή η προσπάθεια, να δούμε ε, τι εντυπώσεις θα, ακούσουμε, θα ακουστούν σύντο χρόνο. Την περασμένη εβδομάδα Ήμουν ε, επικεφαλής ε, μια πολύ ισχυρή αντιπροσωπείας ε, της Επιτροπής μας. Ήταν και η, η Εύλιν Γκέπχαρτ μαζί, που είναι η μόνη που είναι εδώ σήμερα από τους συναδέλφους που ήταν εκεί, για μια πολύ επικοδομητική και νομίζω πολύ σημαντική επίσκεψη στην Κίνα και στο Χονγκ Κόνγκ και ειδικότερα για να επικεντρωθούμε σε ορισμένα ζητήματα που είναι σημαντικά για μας, ε, συγκεκριμένα σε σχέση με την ασφάλεια των προϊόντων των ε, καταναλωτικών. Η κυρία, Μπέγχα, κυρία Γεπχαρτ ε, ασχολήθηκε με πολλά ζητήματα που αφορούν την προστασία των καταναλωτών στην Κίνα. Υπάρχει ένας νέος νόμος όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών στο ίντερνετ και τις δημόσιες συμβεβάσεις. Όταν ήμασταν στο Χονγκ Κόνγκ είχαμε πολύ σημαντικές ανταλλαγές απόψεων όσον όσον αφορά ε, την ασφάλεια της, ε, των πληροφοριών και των ε, δικτύων ε, είχαμε πάρα πολύ λεπτομερές συνεδριάσεις με τους εταίρους μας εκεί για τις μελλοντικέ πολιτικές που θα ακολουθήσουμε και ελπίζουμε ότι το αρμόδιο συμβούλιο στην Κίνα ε, αυτή τη βδομάδα θα ανακοινώσει ένα νέο οικονομικό σχέδιο που θα επικεντρωθεί περισσότερο σε καταναλωτικά προϊόντα και θα συνεχίσει τις ε, μεταρρυθμίσεις της αγοράς. Είχαμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό σημαντικές συζητήσεις όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες και τις φιλοδοξίες της Κίνας προκειμένου να κάνει μια νέα προσφορά ε, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας για τις δημόσιες προμήθειες ε, στον ΠΟΕ. Είχαμε και με τον Επίτροπο πολλά, ζητήματα για την, πολλές ε, συζητήσεις για τα ζητήματα που αφορούν την, τις άδειες για τις εξαγωγές. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η επίσκεψη αυτή και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή την επίσκεψη με τόση ενέργεια και τόσο ζήλο. Στο επόμενο ενημερωτικό μας φυλάδιο θα συμπεριληφθούν όλα αυτά για να μπορείτε να τα δείτε με περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχουν άλλα σχόλια προς αυτά που είπα? Όχι, ωραία. Υπάρχουν τα πρακτικά της 25ης-26ης Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου 2013 θα ε, θεωρηθούν εγκεκριμένα αν μέχρι το τέλος της Επιτροπής δεν γύρει κανείς αντιρρήσεις. Ωραία. Περνάμε λοιπόν τώρα στην πρώτη μας νομοθετική συζήτηση για σήμερα, που είναι η γνωμοδότησή μας για τα δικαιώματα των ε, επιβατών αεροπορικών εταιριών. Να δώσουμε μεγάλη χαρά στον Hans Peter Mayer τον ε, συντάκτη γνωμοδότησή μα, και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Βέστφαλε, Ροσφόρ, Ρούλε, δεν ξέρω αν είστε σκιώδη εισηγήτρια, αλλά νομίζω ότι θα είναι και η κυρία Σούρο, ο κύριο Μπίλεν που δεν είναι εδώ και ο κύριο Ντεγιόγκ, ο οποίο δυστυχώ δεν θα μπορεί να είναι παρόν και οποιοδήποτε άλλο βέβαια θέλει να πάρει το λόγο. Πρόκειται για γνωμοδότησή μας στην Επιτροπή Μεταφορών. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και τις συμβαστικές τροπολογίες. Hans Peter. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μια γνωμοδότηση μεν προς την Επιτροπή Μεταφορών. Πλην όμως έχουμε ασχοληθεί και εμείς εντατικά με αυτό το θέμα όχι μόνο οι δύο αυτές επιτροπές, αλλά και ε, πολύ εντατικά έχουν εργαστεί ο εισηγητής με τους σκιώδεις εισηγητές. Οπότε είμαστε σε θέση πλέον να ε, προτείνουμε συμβαστικές προτάσεις, εννέα τον αριθμό, από 237 ε, συνολικά τροπολογίες. Βέβαια, Απομένουν και ορισμένε που θα πρέπει να ψηφίσουμε, γιατί δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε. Αλλά νομίζω σε κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα κάπου τα βρήκαμε έτσι. Καταλήξαμε σε ένα λογικό αποτέλεσμα. Καταρχάς θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται για τα δικαιώματα των επιβατών των ε, αεροπλάνων και όχι για τα δικαιώματα των αερομεταφορέων και τα οικονομικά των εταιριών. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Μπορεί να παίζουν ρόλο και τα σκεφτόμαστε, αλλά στο προσκήνιο είναι επιβάτης για μας. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν κάνει προτάσεις και ξέρω ότι δεν τους ικανοποιούν ιδιαίτερα ούτε οι τροπολογίες μας ούτε οι συμβαστικές. Κάτι που με ενοχλεί ιδιαίτερα μέχρι που με εκνευρίζει είναι ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείε λένε «Ε, δεν πειράζει τότε θα ε, ακυρώνουμε τις πτήσεις, δεν θα πετάμε καθόλου. Και ε, επανειλημμένα και σε έντονο ύφο έχω πει ότι δεν μπορώ να τα ακούω πια γιατί μας απειλούν ότι θα παρανομήσουν. Μα δεν μπορεί κανείς να ε, μας απειλεί ότι αν δεν περάσει το δικό μας θα παραβούμε μια συνθήκη που έχουμε υπογράψει μια σύμβαση. Δεν επιτρέπονται αυτά. Εκατοντάδες email κυριολεκτικά μας έχουν ε, κατακλείσει μέχρι και σήμερα. Τα έχετε λάβει και εσείς φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπονται και θα πρέπει να ε, τεθεί ένα τέρμα σε όλη αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, να μπω στις συμβαστικές τροπολογίες σύντομα και μετά αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε επί της ουσίας. Συμβιβαστική παριθμών 1 Μιλάει για έκτακτες περιστάσεις. Τι είναι αυτές οι έκτακτες περιστάσεις. Είναι ένας ανοιχτός κατάλογος στο παράρτημα, όχι εξαντλητικός. Είναι αυτές που γίνονται δεκτές και ποιες δεν γίνονται δεκτές από τις περιστάσεις αυτές, τις εξαιρετικές και τις έκτακτες. Υπάρχει μια νομική ε, υπόθεση εδώ θα πρέπει να αποφασίσουμε ποια νομικά οδηγούν σε αποκλεισμό και ποια όχι, αλλά δεν μπορούμε σήμερα να το αποφασίσουμε. Μπορεί να συμβεί κάτι έκτακτο που δεν μπορούσαμε να το έχουμε λάβει υπόψη μας γιατί δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν και δεν θα πρέπει ο κατάλογος, επαναλαμβάνω, να είναι εξαντλητικός. Αλλά ούτε να αφήνουμε στη διακριτική ευχαίρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το συμπληρώνει, αλλά συμμετέχουμε και με τις κατεξουδότηση πράξεις και να ελέγχουμε αν μπορούμε να το επιτρέψουμε ή όχι. Συμβασμός υπαριθμών 2. Αυτό είναι πάρα πολύ επίμαχο σημείο. πολιτική no-show και πάρα πολύ κρίσιμο. Θα σας πω τι είναι αυτό. Οι αεροπορικές εταιρείες θέλουν να διατηρήσουν αυτά που ισχύουν τώρα. Το καταλαβαίνω από τη σκοπιά τους αν θέλετε. Ο συμβιβασμός όμως προτείνει το εξής. Ένας επιβάτης που αγόρασε και πλήρωσε ένα εισιτήριο δεν μπορεί να χάσει όλο το εισιτήριο εάν δεν ε, ε, κάνει τη μία διαδρομή. Έχει πληρώσει ολόκληρο το εισιτήριο. Όταν το εισιτήριο αποτελείται από περισσότερες διαδρομές και δεν έχει πετάξει ας πούμε, τη, μία διαδρομή, γιατί δεν μπορεί να κάνει τις υπόλοιπε. Και με τις σημερινές τεχνικές δυνατότητες δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το αποκλείουν οι εταιρείε. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά επιχειρήματα από πλευρά επιχειρηματικής ε, και υπολογισμούς εταιριών τα κατανοώ. Δηλαδή όταν δεν εμφανιστείς για μια πτήση μου τρως μια θέση και θα μπορούσα να την έχω ξαναπουλήσει. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά την έχει πληρώσει ε, ο επιβάτης και ε, το υπόλοιπο που έχει πληρώσει θα πρέπει να μπορεί να ταξιδεύει. Συμβιβασ ειδική τρία έχει να κάνει με την καθυστέρηση ε, στο διάδρομο ε, στο έδαφος ε, από πέντε ώρες που πρότεινε στην αρχή έχουμε φτάσει στις τρεις ώρες. Το καταλαβαίνω, είναι θέματα του καιρού, έρχεται ο χειμώνας, πρέπει να την χάνουν κάποιες επεξεργασίες ε, με αντιψυκτικά υγρά τα αεροπλάνα, καθυστερούν, μετά προσγειώνεται, πρέπει ξανά να το ψεκάσουν, αλλά μιλάμε για δύο ώρες μέσα στο αεροπλάνο και στο ε, διάδρομο, στο έδαφος, στο αεροδρόμιο για δύο ώρες. Τώρα θα πρέπει λίγο να τα βρουν τους πιλότες, πιλότους οι εταιρείε, δηλαδή δύο ε, ώρες είναι το αεροπλάνο και περιμένει αν είναι 2 και 5 ή 2 και 10 μετά τι θα πει ο πιλότος ότι όχι γυρίζω πίσω ενώ είμαι δεύτερος ή τρίτος στη σειρά για απογείωση α, έχει περάσει το 2ωρο ε, ακύρωση της πτήσης στο 4 η, η διανυκτερεύση σε ξενοδοχεία ε, σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης ή ε, ε, σε περίπτωση που δεν ε, φταίει ο επιβάτης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 100 ευρώ maximum ε, τρεις διανυκτερεύσεις. Οι τροπολογίες ζητούν 100 ευρώ μέχρι 250 ευρώ ή και ορισμένοι το αφήνουν ανοιχτό όσα έξοδα έχει ο επιβάτης. Και επίσης στις τροπολογίες ζητούν ορισμένοι από 0 ε, διανυκτερεύσεις μέχρι άπειρο. Εντάξει, δεν γίνεται εκεί συμβιβασμός. Λοιπόν, εμείς τώρα προτείνουμε 175 ευρώ και περιορισμό των διανυκτερεύσεων σε 5. Συμβαστική παριθμό 5. Η πολιτική ενημέρωση όταν έχει καθυστέρηση πτήση. Το συντομότερο θα πρέπει να δίδεται η ενημέρωση αυτή στους επιβάτες. Ανεξαρτήτως ε, ε, κάποιων στοιχείων που σας στέλνονται στο κινητό τηλέφωνο που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, δεν έχουν όλοι κινητό. Δεύτερον, πριν μπουν στο αεροπλάνο, ο κόσμος το κλείνει το κινητό του, γιατί πρέπει να το κλείνει. Οπότε πώς θα ενημερώνεται. Ε, άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι υποχρεωμένες οι εταιρείε να ενημερώνουν. Σήμερα υπάρχουν τεχνικές τέτοιες δυνατότητες και δεν τίθεται κανένα θέμα. Συμβασμός υπαριθμών 6. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλεγε το άρθρο 16α για τις απαιτήσει και τα παράπονα των επιβατών. Είναι λίγο συγκεχημένη η διατύπωση εκεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα γερμανικά ε, τις απαιτήσει και τα παράπονα. Γιατί ε, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τι εστί απέτηση, τι εστί παράπονο. Είναι νόμος αυτό που ε, προετοιμάζουμε και δεν θα πρέπει να καταλήξουμε στα δικαστήρια. Απέτηση σημαίνει ότι θέλω ως επιβάτης να αποκομίσω κάτι ε, κατά αποκοπή αποζημίωση ή έχω μια απέτηση απέναντι στην εταιρεία. Το παράπονο ή καταγγελία δεν σημαίνει ότι ζητάω κάτι, αλλά κάτι με έχει εκνευρίσει. Ε, η γλώσσα, ο τρόπος που μου φέρονται, η συμπεριφορά ή η άγνοια ή η... καμία ε, πληροφόρηση. Θέλω κάπου να μπορώ να κάνω τα παράπονά μου. Δεν σημαίνει ότι έχω πάντα απέτηση χρηματική ή άλλη. Συμβιβασμός 7 αποσκευές και ενημέρωση για ενδεχόμενα τέλη που θα πρέπει να καταβληθούν. Αυτό θα πρέπει να είναι σαφές από την αρχή, ε, δηλαδή από τη στιγμή που αρχίζει η κράτηση του εισιτήριου και όχι στο τέλος. Ε, και επιπλέον ε, ορισμένα τέλη ενδεχομένως να μην υπάρχουν κάποια κρυφά τέλη που έρχονται να προσθεθούν για τις βαλίτσες στο τέλος. Παράδειγμα, Ε, ε, κλείνεις το εισιτήριό σου, το πληρώνεις ε, και ε, σου λέει «Α, πληρώνεις με πιστοτική κάρτα, συν 20 ευρώ τέλη ε, χρήση πιστοτικής κάρτας». Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, θα πρέπει από την αρχή να είναι γνωστή η ε, συνολική τιμή. Συμβιβαστική 8, απαραίτητα προσωπικά είδη και αγορές από το αεροδρόμιο. Και εκεί υπάρχουν κάποια όρια που θα πρέπει να τα ορίσουμε. Στη Lufthansa, ας πούμε, η χειραποσκευή είναι 55 επί 43, δεν θυμάμαι τώρα πόσα εκατοστά, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Αν αγοράσεις κάτι έξτρα, δεν το μετράς με τον όγκο πλέον, γιατί ο ένας αγοράζει ένα μπουκάλι κρασί και όλος δεν ξέρω εγώ τι. Ε, δεν γίνεται με τις διαστάσεις, αλλά με το βάρος. Ας πούμε, συν 5 κιλά και το σηκώνουν τα αεροπλάνα, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Και πολύ γρήγορα μπορείς και να το ζυγίσεις το check-in, να ξέρεις αν είσαι στα 5 κιλά ή αν τα ξεπερνάς. Δεν χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις στα αεροδρόμια. Συμβασμός 9, 28 ημέρες ε, παράταση της προθεσμίας για ή, μάλλον συντονισμό. Δεν έχουν όλοι τι ίδιε προθεσμίε. Καλό είναι να τι συμπλησιάσουμε για τι διάφορε πληροφορίε. Για την καθυστέρηση, νομίζω για τι 3 και 5 ώρε έχουμε συμφωνήσει μέχρι 3.500 χιλιόμετρα. Τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται με τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, της ε, υπερπόντιες ε, από τη μια είναι Ευρώπη, από την άλλη είναι πολύ μακριά όμως. Οπότε εκεί αντί για τρει ώρε θα μπορούσε κανεί να προτείνει τι πέντε. Είμαι πρόθυμο να το συζητήσω, δεν είναι τραγικό αυτό για μένα. Αυτά, σύντομη παρουσίαση από πλευρά μου. Θέλουμε να συζητήσουμε περισσότερο παρά να αγορεύω εγώ. Οι σκιώδει ηγητέ τα ξέρουν όλα αυτά. Τα έχουν έτσι κάπω χωνέψει και με πολλέ νομοδοτήσει έχουν δώσει τη δική του άποψη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Uh, Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή των συμβαστικών τροπολογιών. Ας δούμε τι λένε οι σκιώδεις, η κυρία Βεσφάλε. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε καθηγητά, κύριε Μάγερ. Στο Στρασβούργο συναντηθήκαμε συνεδρίαση των σκιωδών ηγητών. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική, ανταλλάξαμε απόψεις, κάναμε και ερωτήσεις, ε, μας απαντήθηκαν και σας διαβεβαιώ ότι και το σχέδιο και οι τροπολογίες που κάναμε όλοι μας βρίσκουν νομίζω σύμφωνος. Η δική μου ομάδα έχει κάνει πάρα πολλές τροπολογίες και στόχος είναι ακριβώς να βελτιωθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως να είναι προς όφελος των καταναλωτών στην Ευρώπη, ε, αδρών και γυναικών και να αποτελέσει πρόοδο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τις περισσότερες τροπολογίες θα τις υπερψηφίσουμε και κυρίως τις συμβιβαστικές, γιατί υπάρχουν ε, πραγματικά ε, σημεία όπου έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση μας, δεν μας ικανοποιούν τα πάντα, αλλά τι να κάνουμε, οι συμβιβασμοί αυτό έχουν, έχει και υποχωρήσεις. Αυτό με τις έκτακτες περιστάσεις δεν ξέρω, μας δυσκολεύει λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Θα το δούμε στα νομοθετήματα και ο αριθμός των ορών. Ήταν διαφορετικέ οι προτάσει. Πρέπει όμω να σα πω ότι υπάρχει ένα θέμα που δεν μπορούμε να το δεχθούμε και θα ψηφίσουμε διαφορετικά, διότι πιστεύω ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η δυνατότητα δηλαδή οι αεροπορικές εταιρείε να κάνουν μία έκτακτη ε, κατηδίαν συμφωνία εταιρείε με του επιβάτε. Ξέρουμε τι είναι έκτακτε περιστάσει. Δηλαδή, Όταν κάποιος ε, σύρεται στο αεροδρόμιο ώρες ολόκληρες, θέλει να πάει σπίτι του, θέλει να μπει σε ένα αεροπλάνο και είναι βάλωτος ο επιβάτης της πιέσης. Ε, ανθρώπινο είναι αυτό, έχει την οικογένειά του, παιδιά και ε, τον πιέζουν οι εταιρείε. Λοιπόν, δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο της εθελούσιας ιδιωτικής συμφωνίας ε, διμερός της εταιρεία με τους επιβάτες, τους μεμονωμένους. Κατά τα άλλα συμφωνούμε πάρα πολύ είναι προ όφελο πραγματικά των καταναλωτών, ανδρών και γυναικών. Αυτοί πετούν στο κάτω-κάτω και δεν μας ενδιαφέρει η μεγιστοποίηση του κέρδους των εταιριών. Γι' αυτό χάρηκα πάρα πολύ. Γι' αυτό που είπατε για την πολιτική no-show. Δεν μας ενδιαφέρει η μεγιστοποίηση του κέρδους των εταιριών. Ούτε αρμόδιοι είμαστε γι' αυτό και σε συνεννόηση με τον κύριο Μπαχ συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά, τον, τον εισηγητή της Επιτροπής Μεταφορών. Ήταν παρόν σε όλες τις συνεδριάσεις και των σκιωδών εισηγητών μας. Συνολικά θέλω να πω ότι τα δικαιώματα των επιβατών είναι κάτι που κάνει το Κοινοβούλιο να δείχνει για μια ακόμα μια φορά ότι αποφασίζουμε για τους επιβάτες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορούν να λυθούν σε εθνικό επίπεδο αυτά τα θέματα ο καθένας ε, στη μικρή του γειτονιά. Και, και είδα ότι και η Λουφθάνσα και οι άλλες εταιρείες έχουν δημιουργήσει μια ειδική υπηρεσία για να μπορεί να απευθύνεται ο καταναλωτής και να τον ενημερώνουν και να τα αποκρίνονται στο καθήκον του με διαφάνεια. Νομίζω ότι πραγματικά είμαστε στο σωστό δρόμο και οι νόμοι είναι καλοί όταν δεν καλείται κάποιος να τους ε, εφαρμόσει υποχρεωτικά. Έχουν και μια προληπτική δράση και αυτό είναι πάντα προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ. Ο κύριος Ροσφό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, καθηγητή Μάγερο, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ε, συνεργάστηκε με τους συναδέλφους του προκειμένου να υπάρξει σύγκληση απόψεων. Πραγματικά όταν βλέπουμε τις συμβαστικές τροπολογίες ε, καταλαβαίνουμε ότι είναι πραγματικά από πρώτο χέρι η εμπειρία των πραγμάτων αυτών που αναφέρει. Είναι βιωμένη η εμπειρία ε, εμείς θα υποστηρίξουμε την ουσία των συμβιβαστικών τροπολογιών. Ε, σας το λέω, δεν είναι λοταρία τα νούμερα που θα πω. Σας λέω τον αριθμό των συμβιβαστικών τροπολογιών. 1, K1, 5, 6, 7 και 9. Αυτός είναι ο αριθμός των τροπολογιών των συμβιβαστικών 1, 4, 5, 6, 7 και 9 είναι αυτές ε, οι ε, τροπολογίες συμβιβαστικέ που εμείς ε, υποστηρίζουμε. Για τις υπόλοιπες δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε θέση ακόμη να τις υποστηρίξουμε. Η πρώτη τροπολογία που μας δημιουργεί πρόβλημα είναι το 2, η τροπολογία 2 που αφορά τη μη εμφάνιση των επιβατών, το no-show. Εμείς εδώ είμαστε για να υπερασπιστούμε τον καταναλωτή, να βοηθήσουμε την οικονομική δραστηριότητα. Δεν θέλουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των αεροπορικών εταιριών, οπότε βρίσκω ότι δεν μπορώ να συμπορευτώ με τέτοιου είδους λογική. Αλλά η συμβαστική τροπολογία που αναφέρεται αυτή τη στιγμή, που αναφέρει απλώς άρνηση επιβίβασης για, για οποιοδήποτε λόγο no-show, μας δημιουργεί πρόβλημα Γι' αυτό θα προτιμούσα μια διατύπωση στην οποία θα λέμε ότι απαγορεύεται να αρνούμαστε την επιβίβαση λόγω no-show αν είναι καλή την οι επιβάτες και αν έχουν έναν καλό λόγο να μην έχουν πάρει την πτήση. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει στις ε, τιμολογιακές πολιτικές ανατμήμα ε, υπάρχει μια λογική πίσω από τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες βέβαια θέλουν να γεμίσουν τα αεροπλάνα τους με χαμηλότερες ε, τιμές, χαμηλότερους λάβρους για όσους θέλουν να πάνε στον προορισμό τους με ανταπόκριση ε, και τους δίνουν έτσι ένα χαμηλότερο ναυλό ε, και έτσι γεμίζουν και τα αεροπλάνα τους. Αν εγκρίνουμε αυτήν την τροπολογία ως έχει, ευνοούμε μία συμπεριφορά η οποία πρόκειται, η οποία... Ε, αφορά έναν ε, καταναλωτή ο οποίος ε, φεύγει από, την, ε, από μια, έναν προορισμό που δεν είναι ο προορισμός στον οποίο μένει και κάνει no-show σε, μια, σε ένα τμήμα της πτήσης Παίρνει όμω την ε, υπόλοιπη διαδρομή, ταξιδεύει την υπόλοιπη διαδρομή, ακριβώ για να αποφεληθεί του χαμηλότερου ναύλου. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτό είναι ε, σωστό εκ μέρου μα, ω νομοθέτε να ακολουθήσουμε αυτή τη λογική. Αν ακολουθήσουμε αυτό το κείμενο θα αυξηθεί ο αριθμός ε, μη εμφάνισης των επιβατών, ε, θα υπάρξει overbooking από τις ε, αεροπορικές εταιρείες για να γεμίζουν τα αεροπλάνα τους και επίσης θα έχουμε κάτι το οποίο ε, ουσιαστικά θα ε, μειώσει την ποιότητα της υπηρεσίας αντί να τη βελτιώνει. Γι' αυτό ακριβώς ε, εγώ αυτή τη συμβαστική τροπολογία δεν μπορώ να την υποστηρίξω. Η συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3 είναι αυτή που αφορά το να παραμένουν τα αεροπλάνα στον αεροδιάδρομο κολλημένα. έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές αυτή την εμπειρία, όπως και ο συντάκτης γνωμοδότησής μας. Δεν υπάρχει όμως η ίδια ευελιξία για τις δύο περιστάσεις που αναφέρονται ε, στην τροπολογία αυτή. Δηλαδή υπάρχει μία ανοχή ως προς το να μην γυρνάει πίσω το αεροπλάνο σε περίπτωση ε, αναχώρησης όταν πρόκειται για επικείμενη ε, απογείωση, όταν πρόκειται δηλαδή για απογείωση θα λάβει χώρα στην επόμενη μισή ώρα ε, όταν όμως ε, πρόκειται για την πρόσβαση σε αναψυκτικά ή στις τουαλέτες ε, για παράδειγμα. Αυτή η ευελιξία έχει άμεση σχέση με την, το κατά πόσο είναι επικείμενη η απογείωση ή όχι. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί κανεί θα διαφωνούσε με τα αναψυκτικά στα αεροπλάνο, αν κάποιο είναι κολλημένο με στα αεροπλάνο. Αν όμω σε 10 λεπτά φύγει το αεροπλάνο, τι θα γίνει. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε την ευελιξία αναλόγως με την περίσταση. Γιατί μπορεί να βρεθούμε σε μία περίπτωση ε, αντίθετη τελικά από αυτή που θέλουμε να πετύχουμε. Δεν είναι καλό να, να ψηφίζουμε κείμενα τα οποία τελικά δεν θα εφαρμοστούν ε, ή θα εφαρμοστούν με τρόπο που δεν μας βρίσκει σύμφωνο. Τέλος πάντων η διατύπωση εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και υπάρχει επίσης και το θέμα της ανοχής ε, για τα, τις επιπλέον αποσκευές ε, εντός του αεροσκάφους. Ξέρετε ότι θέλουμε τα duty free να μπορούν, τα ψώνια duty free να μπορούν ε, να τα πάρουν τη στιγμή εκείνη που θα μπαίνουν στο αεροπλάνο μαζί τους χωρίς να θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στο μέγιστο αριθμό αποσκευών ε, που τους επιτρέπεται να βάλουν στο αεροσκάφος. Ε, η συμβαστική τροπολογία αυτή κατά την άποψή μου οδηγεί σε κάτι που δεν είναι ε, σαφές. Γιατί νομίζω ότι τα βασικά αντικείμενα που μπορεί να θέλει να αγοράσει κάποιος ας πούμε από το duty free, μάλλον τα έχει βάλει στις αποσκευές του που θα τα πάρει μαζί, θα τα μαζί του ή άλλως. Οπότε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό, γιατί προσθέτουμε το duty free ε, ε και θέλουμε να το συμπεριλάβουμε στις ε, χειραποσκευές. Για μένα δεν μου φαίνεται δικαιολογημένο αυτό. Εντάξει, είναι σημαντικό, σημαντική πρόθεση για αυτά τα απαραίτητα προσωπικά αντικείμενα, εν πάση περιπτώσει, αλλά πρέπει να ορίσουμε τι ακριβώς είναι αυτά τα ε, αντικείμενα και τι θα μπορεί να παίρνει μαζί του τελικά ε, στην καμπίνα του αεροσκάφους ο επιβάτης. Αυτά ε, είναι τα στοιχεία για τα οποία δεν είμαστε απολύτως σύμφωνοι. Για τα υπόλοιπα συμφωνούμε απολύτως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κείμενο, βελτιώνει την κατάσταση ε, για ένα πρόβλημα το οποίο σημαίνει βέβαια τεράστια ταλαιπωρία και για τους καταναλωτές αλλά και για τον κλάδο γιατί πολλές φορές ε, ε, επαγγελματικά συνέδρια διακόπτονται ή αναστατώνονται λόγω τεράστιων καθυστερήσεων, τουλάχιστον αποζημιώνεται ο κόσμος Αυτά λοιπόν ήθελα να πω εκ μέρου τη ομάδα μας για τις συμβαστικέ τροπολογίες του κυρίου Μάγερ. Ευχαριστώ. Uh, thank you very... Σας ευχαριστώ. Ίσως ε, δεχθήκαμε λίγο αργά το σχέδιο κάποιων τροπολογιών. Ε, κυρία ε, Σούλα. Κυρία Ρούλε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, συμφωνούμε με τους συμβιβασμούς, τους υποστηρίζουμε και σε αντίθεση με τον προλαλήσαντα θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι αυτή η αρχή της μη εμφάνισή του no-show, είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι σοβαρές οι εταιρείε, κάνουν αυτούς τους υπολογισμούς και τη σπέκουλα και ε, ε, έχει πληρώσει ο επιβάτης και θα πρέπει να τον ενημερώνουν. Εάν κάνει διαφορετικό υπολογισμό η εταιρεία να τον αλλάξει. Μπορεί να είναι πιο ακριβή η πτήση, αλλά αν υπάρχει διαφάνεια μπορώ να το δεχτώ. Αυτά, πάντα υπέρ της διαφάνειας. Um, λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει με τους κοιόδης. Ε, η η κυρία Στάιλερ έχει ζητήσει το λόγο. Δεν ξέρω αν κάποιο άλλο μέλος θα ήθελε το λόγο. Ή μήπως κάποιος από την Επιτροπή που ήθελε να μιλήσει. Συγγνώμη, δεν σας είδα, λέει ο Πρόεδρος. Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο αμέσως μετά. Η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους και ε, Νομίζω ότι είχαμε εξαιρετική συνεργασία και κρίμα που δεν έχουμε και περισσότερους φακέλους ε, με τόσο καλή συνεργασία. Για τις συμβαστικές, ε, πολύ χαίρομαι που φτάσαμε στο όριο των δύο ωρών. Είναι ενθαρρυντικό. Άκουσα και τον ε, σκιώδη συγητή, την σκιώδη συγητή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών σχετικά με το εθελούσιο του ορίου αυτό. Πρέπει να είμαστε δεσμευτικοί σε αυτά που κάνουμε. Γιατί όπως είχα πει ε, πρέπει να βλέπουμε ε, αυτά τα σημεία ως παραδείγματα βελτίστων πρακτικών και χειρίστων πρακτικών των αεροπορικών εταιριών μερικές φορές. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πρακτικοί για να μπορέσουμε να βρούμε μια σωστή λύση και να έχουμε σωστή προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Τώρα σχετικά για το χρονισμό, στην άλλη επιτροπή ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή, γιατί φτάνουμε στο τέλος της εντολής, ήθελα να καταλάβω με το χρονισμό πώς θα πάμε με αυτό το φάκελο, αλλά νομίζω ότι η συνεργασία που έχουμε δει με τις άλλες επιτροπές με στιγμή ε, θα πρέπει να την επαναλάβουμε και στο μέλλον και θα πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε ως πρότυπο, ως παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ επιτροπών, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος. Παρακαλώ. Ας ακούσουμε από την Επιτροπή. Δεν είχα το όνομά σας στον κατάλογό μου, ζητώ συγγνώμη. Από την ε, γάμα δελτα μουβ είναι το μόνο που ξέρουμε. Ναι, καλησπέρα σας Ντανιέλα Κίτη από την ε, Digimove. Ασχολούμαστε με τα δικαιώματα των ταξιδευτών ε, έχοντας ακούσει τώρα τον εισηγητή και τους εσκαιώδεις εισηγητές που τοποθετήθηκαν από πλευρά τη Επιτροπή, ε, μπορούμε να σας πούμε ότι χαιρόμαστε που κάποιες από τι συμβαστικέ τροπολογίε ε, πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, διαφημίζουν κάποια δικαιώματα σχετικά με την πολιτική με εμφάνιση. Για παράδειγμα, είχαμε υποστηρίξει απολύτω. Από την άλλη μεριά, θα ήθελα να σημειώσετε ότι μερικές φορές οι καταναλωτές, οι ταξιδιώτες, και αυτό το είχαμε σημειώσει ο πλευράς επιτροπής, πολύ συχνά ενώ η συμφωνία φαίνεται καλή στο χαρτί, έχουμε έμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην πράξη. Και εδώ σκέφτομαι την ε, πρόταση νέου δρομολογίου σε περίπτωση καθυστέρηση. Αυτό δεν αναφέρθηκε εδώ, αλλά σας δίνω ένα παράδειγμα. Αν, επί παραδείγματι, ε, προτείνουμε μετά από δύο ώρες καθυστέρηση νέα διαδρομή, νέο δρομολόγιο, αυτό θα είναι κατά των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Μερικές, ε, μερικοί μεταφορείς δεν έχουν καν εναλλακτική λύση να προσφέρουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και ο επιβάτης ε, αναγκάζεται να ακολουθήσει νέο δρομολόγιο και να έχει καθυστέρηση ε, μερικές φορές άραν των 12 ωρών. Και να υπογραμμίσω και μία άλλη πτυχή. Έχουμε μία ιδεολογική σκέψη αυτή τη στιγμή στον κανονισμό και προσβλέπουμε στην προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Θέλουμε να έχουν ασφαλές ταξίδι, αλλά εξετάζω τις τροπολογίες σχετικά με τις έκτακτες συνθήκες. Αυτός ο μη εξαντλητικός κατάλογος. Γιατί είμαστε υπέρ του μη εξαντλητικού καταλόγου από πλευρά τη Επιτροπή. Όπω είπε και ο εισηγητή, υπάρχουν εξορισμού περιπτώσει που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Και υπάρχουν περιπτώσει που δεν μπορούμε να τι περιγράψουμε που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τέτοιε συνθήκε. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ποια στοιχεία αυτός ο κατάλογος θα συμπεριλαμβάνει, διότι πρέπει να διατηρούμε υπόψη μας τα μέτρα ασφαλείας. Και όπως έλεγα αυτό που επιθυμούμε εμείς από τον κανονισμό αυτόν είναι να παράσχει το πλαίσιο ασφαλούς ταξιδιού για τους επιβάτες. Να μην δίνει κίνητρα δηλαδή ούτε ακύρωσης για τους αερομεταφορείς, ούτε να εκτελείται η πτήση από κατά που να μην είναι ασφαλής. Αυτά είναι τα βασικά σχόλια, ίσως κάτι τελευταίο από πλευρές Επιτροπής. Ήθελα να θυμίσω στα μέλη την πρόθεση της Επιτροπής, η οποία ήταν σχετικά με την παραμονή των επιβατών, τη διαμονή τους, όχι μόνο για να άρουμε λίγο από το άχθος επί των αερομεταφορέων, αλλά και για να ευθυγραμμίσουμε τις διατάξεις αυτές με άλλες, με άλλα νομοθετήματα που προέβλεπαν διαμονή για τους επιβάτες ε, στο πλαίσιο των μεταφορών και έχουμε και τα σχέδια δράσεως τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε για τέτοιες περιπτώσεις για να προστατεύονται τα συμφέροντα των επιβατών και για να αποφεύγονται δυσάρεστες εκπλήξεις, ας πούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ που μας δώσατε την οπτική της Επιτροπής. Να δώσω λοιπόν το λόγο ξανά στον κύριο Μάια για να συνοψίσει και να πάμε ε, σε ψήφο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους αγαπητούς συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις συμπληρώσεις της και για τις παρατηρήσεις αυτές. Για τις εθελούς συμφωνίες θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι αύριο ακόμα. Είναι γεγονός. Ε, με την Επιτροπή Μεταφορών. Πώς έχει το διάγραμμα. Σε ένα τέταρτο θα αρχίσει η δική του συζήτηση. Θα πάω κι εγώ εκεί και θα προσπαθήσω να πάρω το λόγο, αν μου το δώσουνε συμφωνούμε σε πολλά σημεία. Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια αριθμητικά στοιχεία, αλλά δεν χάλασε και ο κόσμος. Γιατί πάντα προσκαλούσαμε τον εισηγητή, τον κύριο Μπαχ, ε, στη συζητήση μας και τα ξέρει. Από την αρχή ε, είχαμε μια ανταλλαγή πολύ καλή. Και να δούμε τι θέλει για την πολιτική ε, της μη εμφάνισης του no Δεν ξέρω ακριβώς τι θέλει. Λέει και ξελέει, το είδαν και άλλοι σκιώδησηγητές, θα τα ξανασυζητήσουμε μαζί του. Κατά τα νομίζω, διαπιστώνω μια ευρύτατη υποστήριξη των κοινών άλλωστε συμβιβαστικών προτάσεων. Για τα ασφαλή ταξίδια που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Είναι αυτονόητο. Ό,τι προτείνουμε και ό,τι αλλάζουμε προφανώς δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος ε, της ασφάλειας, ούτε επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι απόφαση της εταιρείας, αλλά τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο έχει ο κυβερνήτης. αν θα ξεκινήσει ή αν δεν θα ξεκινήσει. Δεν έχει καμία σχέση με τον νόμο η ασφάλεια. Μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα ε, τεχνικό στο αεροσκάφος και θα πρέπει να είναι τελείως ανεπηρέαστη η απόφαση. Και η Ένωση ε, των Κυβερνητών ε, Πιλότων που είναι στους θαλάμους διακυβέρνησης το λέγουν, δεν λαμβάνουν υπόψη ποτέ ούτε τις πιέσεις των εταιριών ούτε των επιβατών παρά μόνο την ασφάλεια. Και αν ε, ένα μικρό σωληνάκι ε, που μεταφέρει νερό από τρία έχει τρυπήσει, ας πούμε, μπορεί να πετάξεις. Αλλά αν ανάψει ένα κόκκινο λαμπάκι στο θάλαμο διακυβέρνησης, ε, ξέρουν οι πιλότοι πότε πρέπει να πετάξουν και πότε όχι. δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς με τις εταιρείες να κάνουν συμφωνίες και με ξενοδοχεία και για αριθμό διανυκτερεύσεων. Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Ε, θα πρέπει να τους εξασφαλίζουν διανυκτέρευση. Σε περίπτωση όμως που δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και καλούνται οι ε, επιβάτες να βρουν μόνοι τους ξενοδοχείο, ε, τότε δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις ε, Προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι όλο δεν πάει χιλιόμετρα να βρει ξενοδοχείο, παίρνει το ξενοδοχείο του αεροδρομίου που ξέρουμε ότι δεν είναι και το φθηνότερο. Αυτά. Κατά τα άλλα σας ευχαριστώ πολύ και πρέπει να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ αυτή τη συνεργασία μας για τη συγκεκριμένη νομοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που κάναμε πρόοδο και μάλιστα σας, μάλιστα σας επένεσαν και για τη δουλειά σας. Ελπίζω να επιβεβαιωθεί αυτός ο έπαινος αύριο. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάτε και στην Επιτροπή Μεταφορών όπου συζητούν την έκθεσή τους. Περνάμε τώρα στην επόμενη γνωμοδότηση, για την οποία κάναμε πολλή δουλειά και την έκθεση πρωτοβουλίας αυτή για τους λογαριασμούς πληρωμών υπό την οπτική γωνία του συμφέροντος των καταναλωτών. Η Evelyn Γκέπχαρτ είναι ε, η εισηγήτριά μας. Ε, ξέρω ότι με την ε, εισηγήτρια της Αρμόδιας Επιτροπής δούλεψα πάρα πολύ σκληρά μαζί. Ο κύριος Φαμπ θα μιλήσει εκ μέρους του ΕΛΚ. Ο κύριος Σμίτ δεν είναι εδώ. Η κυρία Ρούλε είναι εδώ. Μιλάει με την κυρία Βάιλερ για την ώρα. Ο κύριος Κούσνικ δεν είναι εδώ. Τέλος πάντων. Απαρτία εισηγητών. Και είναι εδώ και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Νάβα, ο οποίος είναι διευθυντής, ο κύριος ε, Μάριο Νάβα. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίασή μας. Θα σας δώσουμε το λόγο μετά τον πρώτο γύρο συζήτησής μας. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην Εύελιν Κέπχαρ να μας παρουσιάσει τις ε, συμβαστικές τροπολογίες. Εύελιν, έχεις το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δικούς μου σκιώδεις συζητητές με τους οποίους συνεργάστηκα πολύ καλά. Είχαμε πολύ ωραίες συνεδριάσεις στο Στρασβούργο και με ορισμένους ε, την περασμένη εβδομάδα στην Κίνα, ακόμα και με τον κύριο Σφάπ, μέχρι και στην Κίνα συζητούσαμε ε, τις συμβιβαστικές αυτές τροπολογίες. Καταθέτω λοιπόν αυτή τη στιγμή 19 τροπολογίες. Προς Θεού δεν θα σας τις διαβάσω όλες τώρα, θα σας τις παρουσιάσω. Ε, κυρίως την προσέγγισή μας να σας περιγράψω, γιατί είναι σημαντική. Δύο-τρία είναι τα σημεία όπου δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε οριστικούς συμβιβασμούς, αλλά μέχρι αύριο που έχουμε την ψηφοφορία θα πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε. φαντάζομαι ο κύριος Φαμπ θα μπορέσει να μου απαντήσει ε, κάποια από τις ερωτήσεις μου για το τι μελή γενέστε. Λοιπόν, έχουμε ένα σημείο που πρέπει να ορίσουμε για το, ε, το βασικό τραπεζικό λογαριασμό και την αλλαγή ε, λογαριασμού και για ποιες τράπεζες πρόκειται, ποιες είναι αυτές οι τράπεζες που θα πρέπει να τον ε, προτείνουν το λογαριασμό αυτό. Και έχω κάνει λοιπόν μια διατύπωση ε, με σαφέστερο ορισμό. Τι εννοώ. είναι τράπεζες που ε, προσφέρουν ε, γενικά τέτοιους λογαριασμούς σε ιδιώτες, σε πελάτες. Τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να μπει αυτό σε τροπολογία. Ε, εγώ θα πρότεινα κάτι, κύριε Σφάμπ, αλλά δεν συμφωνεί απολύτως η πολιτική σας ομάδα, να το γράψουμε στο άρθρο 2. Ένα ορισμό που να βρίσκει γενική εφαρμογή για όλο το κείμενο. Κατά την άποψή μου αυτό θα είχε μεγαλύτερο νόημα και θα ε, ελάφρυνε γενικότερα ε, όλη την προσπάθεια, καθώς επίσης και την αυριανή ψηφοφορία. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσω την άποψή σας σχετικά. Τώρα, για την αλλαγή ε, λογαριασμού πληρωμών, το λεγόμενο switching, πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να μπορείς να αλλάζεις τράπεζα από χώρα σε χώρα. Ε, πολιτικές ομάδες δεν συμφωνούν σε αυτό όλες. Εγώ συμφωνώ μεν με τη Κομισιόν, αλλά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα νομίζω ε, θέλει περιορισμό. Ότι να μπορεί κανείς να αλλάζει λογαριασμό η τράπεζα στο εσωτερικό της χώρας του. Εντάξει, δεν είναι ευρωπαϊκή υπόθεση αυτή, γι' αυτό το έχω προτείνει ως συμβιβαστική πρόταση. και να έχουμε μία προσέγγιση σε δύο χρόνους. Δηλαδή, να πούμε ότι να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός και από τη στιγμή της θέσεως ισχύ ε, να μπορεί κανείς να αλλάζει λογαριασμό εντός του χώρου ΣΕΠΑ και μετά από μία πενταετία να δούμε ε, αν μπορεί να μεταφέρει το λογαριασμό του ε, σε τράπεζα εκτός χώρου ΣΕΠΑ. Ξέρω ότι θα δυσκολέψουν λίγο τα πράγματα τότε, γιατί υπάρχει και η δυνατότητα και η ανάγκη μετά ε, υπολογισμού των ισοτιμιών κτλ. Άκουσα ότι είχαμε συμφωνήσει, τώρα ακούω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν τα βλέπει ακριβώς έτσι. Κύριε Σουάπ, μπορείτε να μου εξηγήσετε που έχει πρόβλημα η ομάδα σας, γιατί δεν το έχω καταλάβει για να μπορέσουμε να έχουμε μια οριστική διατύπωση μέχρι αύριο για την ψηφοφορία. Και να προσπαθήσω να ικανοποιήσω όλες τις πολιτικές ομάδες γιατί είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν για τη μεταφορά η αλλαγή λογαριασμού, σε άλλη τράπεζα δηλαδή. Τώρα, για την ενημέρωση ε, περί των τραπεζικών τελών, τα έχουμε βρει, δεν χρειάζεται να μπω ε, σε λεπτομέρειες είχαμε συμφωνήσει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει σωστή πληροφόρηση, εύληπτη, κατανοητή και προσβάσιμη για τους πολίτες ε, όλους, άνδρες και γυναίκες. Δεν διαφωνούμε και δεν θέλω να επεκταθώ. Το ίδιο ισχύει και για τη συγκρισιμότητα των διαφόρων ιστοσελίδων, των τραπεζών κτλ. Μεγάλη σημασία αυτό. Τώρα, σε αυτή την πρόσβαση στο βασικό τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών για πολίτες που δεν έχουν συνήθως πρόσβαση. Και ξέρουμε ότι είναι εκατομμύρια εκείνοι που δεν δικαιούνται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα επιθυμούσαν με να έχουν τραπεζικό λογαριασμό, αλλά δεν τους ανοίγουν οι τράπεζες. Γι' αυτό, αυτό θέλουμε εμείς να επιτύχουμε. να Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν υπάρχει εδώ μεγάλη διαφωνία, ε, όπως σας είπα, με εξαίρεση το εξή σημείο. πώς να το πω, Πώς το λένε αυτό στα γερμανικά. Features. Α, στοιχεία. Ε, αυτό είναι όταν τα συζητάμε στα αγγλικά, ξεχνάμε και τη γλώσσα μας. Ακόμα και οι Γερμανοί στα αγγλικά τα συζητάμε μεταξύ μας αυτά. Λοιπόν, τα διάφορα στοιχεία και ε, θα πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν τι θα προσφέρει αυτός ο τραπεζικός λογαριασμός και πώς θα εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα. Εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 80% των στοιχείων. Ε, αλλά δεν ορίζει ξεκάθαρα τη βάση ε, επί των οποίων προτείνει το 80%. Εγώ θα πρότεινα 90, άλλος θα σου πει 60, Ωραία. Κολοκυθιά. Ε, ο καθένας παίρνει υπόψη του αυτό που λέει η χώρα του. Αλλά τώρα είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και καλό θα ήταν ε, να μπει και το ευρωπαϊκό επίπεδο στο παιχνίδι για να υπάρχει ακριβώ αυτή η δυνατότητα σύγκρισης. Προτείνω λοιπόν να υιοθετήσουμε αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 80% για ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ στα κράτη-μέλη είναι 90% των κοινών στοιχείων που προτείνει κάθε τράπεζα στο λογαριασμό αυτό. Και στο ΕΛΚ ερωτηματικό έχω. Επιμένετε στο 90%? Και πάλι θα μπορούσε να μου απαντήσει εδώ ο κύριος Φαπ. Τι λέει η ομάδα του. Εγώ έχω κάνει μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνσή σας, διότι πάντα θεωρούσα ότι θα πρέπει να ε, υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης όλων των στοιχείων, δηλαδή του 100%. Ε, Παρ' όλα αυτά είμαι πρόθυμη να δείξω μια ευελιξία για να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβιβαστικό κείμενο που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αυτά τα βασικά ερωτήματα. Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα που είχαμε ακόμα να συζητήσουμε. Και τώρα με τεράστιο ενδιαφέρον περιμένω να ακούσω τι θα πούν οι σκιώδεις ή εκπρόσωποι τους. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα αλλαγής λογαριασμού, μεταφοράς του λογαριασμού από μια τράπεζα σε μια άλλη, να είναι απλή αυτή η διαδικασία όσο γίνεται πιο ε, φτηνή για τους πολίτες και η πρόσβαση σε ένα λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να είναι δεδομένη. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά στοιχεία της ευρωπαϊκής πρότασης και να είναι όσο γίνεται πιο απλό για τους πολίτες αυτούς που σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν λογαριασμό. Διότι αυτό που δεν επιθυμώ να δω είναι κάποιοι νέοι ε, που βγαίνουν με εράσμους σε μία χώρα να έχουν βιώματα τελείως αντιευρωπαϊκά. Δηλαδή φτάνουν σε μια χώρα, θέλουν να ανοίξουν λογαριασμό. Ε, μάλλον θέλουν να υπογράψουν ένα συμβόλαιο για να νοικιάσουν σπίτι και σου λέει δεν γίνεται, πρέπει να έχει λογαριασμό στη χώρα. Πάνε στην τράπεζα και λένε Α, δεν γίνεται, άμα δεν έχει διεύθυνση, πώ θα ανοίξει λογαριασμό και να μου φέρει το συμβόλαιο, το νοικιαστήριο. Εγώ δεν θέλω οι νέοι μας να ζουν τέτοια πράγματα στην Ευρώπη και θέλω ε, να τους διευκολύνουμε όσο γίνεται. Αυτό είναι άλλωστε ο στόχος της φέρους νομοθεσίας και χαίρομαι που καταφέραμε με αυτή την έκθεση πρωτοβουλία και νομοθετική να κινήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει και αυτή τούτο το βήμα. Γιατί στην αρχή ήταν μάλλον απρόθυμη. Είναι σημαντικό όμως αυτό για τους πολίτες μας πάντα, άνδρες και γυναίκες. Good. Thank you very much. ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ας ακούσουμε τους ε, σκιώδεις ε, εισηγητές, ο κύριος Σουμπάμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκέμπχαρτ αλλά και εσάς και τους άλλους συναδέλφους για τις επικοδομητικές συνομιλίες και για αυτό εδώ το θέμα. Τα είπαμε μέχρι και στην Κίνα. Αυτά συζητούσαμε. Θα αρχίσω με τα δικά μου σχόλια και μετά θα απαντήσω. Και στα γερμανικά <laughs> να μην, να μην έχουμε προβλήματα γλωσσικά. Λοιπόν, είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας που με πολύ μεγάλη πλειοψηφία τελικά υπερψήφισε η Επιτροπή μας είναι ένα σημαντικό στοιχείο και μήνυμα ακριβώς προς την εσωτερική αγορά και ένα μήνυμα για τους νέους, όχι μόνο τους φοιτητές, αλλά και άλλους. Θυμάμαι όταν, ε, αγαπητέ Μάλκομ, σπούδαζα στη Μεγάλη Βρετανία, μπορούσε κάποιος όταν είχε υποτροφία να ανοίξει δωρεάν λογαριασμό τραπεζικό που σήμερα έχει καταργηθεί, ε, αλλά οι άλλοι που δεν είχαν υποτροφία πρέπει να πληρώνουν και 50 με 60 λίρες το μήνα ως έξοδα τραπεζικά για να έχουν λογαριασμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και ε, χαίρομαι. Είναι μια επιτυχία αυτή που έχει να κάνει και με την καθημερινότητα των πολιτών, την πραγματικότητά τους, ζουν την Ευρώπη στο πετσί τους. Ε, γι' αυτό υποστηρίζω ρητά αυτή την πρωτοβουλία. Είπαμε ήδη ότι ως Κοινοβούλιο το είχαμε ζητήσει αυτό ως έκθεση πρωτοβουλίας και ερχόμαστε στη νομοθεσία για να πάρει σάρκα και οστά. Ελπίζω κυρία Κέπχαρτ αυτά που εκκρεμούν ακόμα τα σημεία να τα βρούμε ε, με επικοδομητικό πνεύμα και συμβιβαστικό. Έχετε δίκιο. Το 80% δεν μας βοηθάει γιατί είναι πολύ συγκεχημένο αυτό στο οποίο αναφέρεται. 80% τίνος. Ποιο είναι το 100% για να καταλάβουμε το 80% που θα ε, εναρμονιστεί, τι θα είναι. Θα το συζητήσουμε. Θα έρθει ο δικός μας και ο το βράδυ και θα ασχοληθεί ο ίδιος με το θέμα. Ε, κατά τα άλλα, κύριε Πρόεδρε, ως αναπληρωτής Κιώδης θα ήθελα να σας εξηγήσω τις θέσεις του κυρίου Μπόρισοφ και όχι του κυρίου Γκέπχαρτ, όπως είπα κατά λάθος, που με παρακάλεσε να σας... Ε, Οπότε εξή. Να ευχαριστήσω την κυρία Γκέφαρτ για την καλή συνεργασία και συνεχίζω στα αγγλικά. Σχετικά ναι. λοιπόν με μια προσέγγιση δύο βημάτων. Με μια προσέγγιση δύο βημάτων σχετικά. Και η διαφορά από αυτά που είπατε κυρία Γκέπχαρτ, μετά από μια μεταβατική περίοδο 5 ετών, να πάμε σε διασυνοριακή λύση. Πρώτα εθνικό βήμα, λοιπόν, <clears throat> και μετά με μια πιο μακριά περίοδο να μπορέσουμε αυτό να το υλοποιήσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, το διασυνοριακό switching, η αλλαγή των λογαριασμών μεταφορά, θα μας ε, επέτρεπε να κάνουμε τις τεχνικές προσαρμογές που χρειάζονται. Διότι στο τέλος έχουμε όλοι το συμφέρον. Οι κάτοχοι των λογαριασμών που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό, αυτό να λειτουργεί και όχι να έχουν εμπόδια, νέα εμπόδια. Επίσης ο κύριος Μπορίσοφ μου ζήτησε να σας πω, σχετικά με την πρόσβαση σε ε, λογαριασμό πληρωμών, θα πρέπει να υπερασπιστούμε μια προσέγγιση ιστορικής αγοράς, επομένως θα πρέπει να πετύχουμε περαιτέρω ενσωμάτωση και να έχουν περισσότερες επιλογές οι καταναλωτές. Είμαστε υπέρ λοιπόν τις δυνατότητες για τους καταναλωτές ανοίγματο βασικού λογαριασμού, βασικών χαρακτηριστικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμβέλειας δηλαδή, που θα είναι ένα ενσωματωμένο κομμάτι, κομμάτι της κανονικής της οικονομικής δραστηριότητας. Για τη συμβαστική πρωτοβουλία επ' αυτού του θέματος είναι υπέρ ο κύριος Μπορίσοφ. Τώρα για τους ε, εργαζομένους, τους αποσπασμένους ή τους μετανάστες θα πρέπει να τροποποιηθούν αντίστοιχα οι διατάξεις. Επίσης σχετικά με τις ονομαστικές αυτές ε, τα τέλη ή όχι, το είχαμε συζητήσει και ο πρόεδρος ο κύριος Χάρμπορ μας βοήθησε ε, με αυτό το nominal, το ονομαστικό που σημαίνει δηλαδή τέλος που βασίζεται στο κόστος στην ουσία. Επίσης για τη διαφάνεια και τον κατάλογο των πιο χρησιμοποιημένων υπηρεσιών, ο κύριος Μπορίσοφ θεωρεί ότι το 80% είναι το καταλληλότερο επίπεδο, αλλά θα πρέπει να δούμε, όπως έλεγα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Δηλαδή ως προς τι 80% και νομίζω ότι επί τη βάση αυτή σίγουρα μπορούμε να βρούμε μια συμβαστική λύση για την αυριανή η ψηφοφορία και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ λέει ο πρόεδρο. Πολύ χαίρομαι που και εγώ μπόρεσα να κάνω μια μικρή συνεισφορά γλωσσικά. Η κυρία Ρούλα. Πολύ σύντομη θα είμαι. Ευχαριστώ την κυρία Γκέπχαρτ για την καλή συνεργασία. Πάντα ε, μας έστειλε τις συμβαστικέ ε, τροπολογίες εγκαίρως. Είχαμε το χρόνο να τις διαβάσουμε γιατί τις υποστηρίζουμε απολύτως. Ευχαριστώ. Okay. Um, to... Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο για τη συζήτησή μας αυτή. Ωραία. Εντάξει. Εγώ θα ήθελα να πω μερικά πράγματα, αλλά μπορώ να τα πω κατευθείαν ε, στον εισηγητή, στην εισηγήτρια, συγγνώμη. Ε, νομίζω ότι συμφωνώ πάντως με τα περισσότερα εξ είπε. Να ζητήσω από τον κύριο Νάβα να σχολιάσει τη δουλειά μας ως τώρα. Πείτε μας ορισμένα πράγματα για το πώς ε, προοδεύει ο φάκελος αυτός. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω καταρχάς την κυρία Γκέπχαρτ και όλους τους κοιόδης εισηγητές ε, γιατί όχι μόνο με καλωσορίζουν εδώ σήμερα αλλά και γιατί έχουν ε, δουλέψει πολύ και αυτό δείχνει πραγματικά ότι και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συμφωνούν ε, για το, στο θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπό είχε με την πρότασή της αυτή να λάβει υπόψη της και όλους όσους, μετακινούνται είτε στο πλαίσιο του Εράσμους, είτε μετανάστες, άνθρωποι, νέοι επιχειρηματίες που δεν έχουν ένα τραπεζικό λογαριασμό και ξέρετε τι θα πει να μην έχει κανείς λογαριασμό, σημαίνει ότι δεν έχει πρόσβαση ε, στην ψηφιακή αγορά σημαίνει ενδεχομένως ότι δεν ε, συμμετέχει πλήρως ε, στην ευρύτερη οικονομία, για να το πω έτσι. Νομίζω ότι τα τρία βασικά ε, θέματα τα αναφέρατε και μπορώ να σας πω ποια είναι η δική μας άποψη. Όσον αφορά την αλλαγή ε, παρόχου υπηρεσιών μας, είπατε ότι μπορεί να είναι πιο εύκολο διασυνοριακά να γίνεται αυτό από ό,τι γίνεται σε επίπεδο εντός ενός κράτους μέλους και ότι θα θέλατε μία λύση γι' αυτό. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαμε δει όντω αυτή τη διαφορά και ενδεχομένως να είχαμε μία διαφορετική λύση προτείνει. Η διασυνοριακή ε, περίπτωση είναι πολύ συνηθισμένη Α σκεφτεί κανεί για παράδειγμα τι διάφορε μεθοριακέ ε, περιοχέ ε, μεταξύ Γαλλία, Γερμανία, ε, Βελγίου, Λουξεμβούργου, Ολλανδία. Υπάρχουν πολλά διασυνοριακά ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ συνηθισμένα, πολύ καθημερινά. Είναι θέμα συνεργασία μεταξύ των τραπεζών, οπότε η αλλαγή από τον έναν τραπεζικό φορέα στον άλλον θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Θέλουμε όμω να δώσουμε πρόσβαση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και όταν έχουν έναν τραπεζικό λογαριασμό δεν θέλουμε να παγιδεύονται σε αυτό γιατί είναι νέοι άνθρωποι, είναι η πρώτη φορά που έχουν έναν τραπεζικό λογαριασμό και μπορεί να μην κάνουν την καλύτερη επιλογή στην αρχή. Πρέπει λοιπόν να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν πάροχο υπηρεσιών τραπεζικών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να βρεθεί ένας τρόπος να μην είναι πιο περίπλοκη η κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα όσον αφορά τη διασυνοριακή αλλαγή υπηρεσιών, όσον αφορά τη διαφάνεια. Καταλαβαίνω ε, τι μας είπατε. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι, εξακολουθεί να ισχύει ακόμα. Ε, και τέλος, όσον αφορά την πρόσβαση που είναι το βασικό στοιχείο, άκουσα την κυρία Γκέπχαρτ να λέει ότι αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας βεβαίως να εξασφαλίσουμε ότι όλοι όσοι θέλουν να έχουν ένα τραπεζικό λογαριασμό να έχουν και Ισχύει και για όσους είναι στο Εράσμους, για παράδειγμα. Αυτοί είναι μάλιστα και πιο προνομιούχοι. Νέοι, φοιτητέ, έχουν όλη τη ζωή μπροστά του. Πολλοί έχουν πάει στο Εράσμου. Ε, είχα και εγώ, όπω και ο κύριο Σφαμπ, μια παρόμοια εμπειρία. Αλλά βλέπουμε και του υπόλοιπου νέου επιχειρηματίε, για παράδειγμα, που θέλουν να ανοίξουν έναν τραπεζικό λογαριασμό και δεν μπορούν να το ανοίξουν τον τραπεζικό λογαριασμό ούτε στη δική τους, ε, στο δικό του τόπο. Ε, λόγω των απαιτήσεων που υπάρχουν. Προσπαθούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε το ότι θα διευκολύνουμε τη διαδικασία όσο δυνατόν περισσότερο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίω θα σα υποστηρίξει και εσά προσπάθειέ σα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τη βελτίωση του κειμένου. Νομίζω ότι κινούνται προ την κατεύθυνση που επιθυμούμε κι εμεί εμείς παραμένουμε δεσμευμένοι στο να ολοκληρωθεί αυτός ο φάκελος συντομότερο δυνατόν, και στο πλαίσιο αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για την ε, πολύ ε, συνοπτική και ενθαρρυντική σας απάντηση. Κυρία Γκέπχαρτ, μήπως θέλετε να συνοψίσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Εσύ ότι μέχρι αύριο θα έχουμε βρει ε, ένα συμβιβασμό που θα μπορέσουν όλοι να συμφωνήσουν, ειδικά ακούγοντα του συναδέλφου, Θα κάνω και εγώ προτάσει προ την κατεύθυνση αυτή, σημειώνοντα τα όσα είπατε. Επιτρέψτε μου όμως να ξεκαθαρίσω το εξή. Ακριβώς η πρόσβαση σε ένα τέτοιο ε, λογαριασμό πληρωμών είναι σημαντική. Και έχετε δίκιο, δεν είναι μόνο οι φοιτητέ που ταξιδεύουν και είχαν αυτή την εμπειρία του Εράσμου. Έχουμε και εποχικούς εργαζομένους. Μικρούς ε, επιχειρηματίες που θέλουν να έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα και χρειάζονται ένα απλό τραπεζικό λογαριασμό για να διεκπεραιώνουν τις ε, εργασίες τους. Πρόκειται όμω επίσης και για αστέγους Φερρυπίν που ε, μαζεύουν κάποια χρήματα και φοβούνται το βράδυ μην τους κλέψουν και δεν κοιμούνται θα προτιμούσαν να τα καταθέτουν σε ένα τραπεζικό λογαριασμό τα λεφτά αυτά που έχουν. Και για αυτούς τους ανθρώπους πρόκειται. Στη σημερινή κοινωνία περίπου δεν θεωρείσαι άνθρωπος αν δεν έχεις τραπεζικό λογαριασμό. Είναι θέμα ανθρώπινης υπόστασης. Das ähm, Αυτά είναι τα σημαντικότερα λοιπόν στη συγκεκριμένη δουλειά που κάνουμε εμείς. Θα ξανακάνω προτάσεις ε, συμβιβαστικές και είμαι βέβαια ότι αύριο θα πάει καλά η ψηφοφορία. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω όλους σας, όλους τους συναδέλφους, γιατί πραγματικά ε, ήμασταν πιεσμένοι χρονικά για να μπορέσουμε εγκαίρως να καταθέσουμε στην ε, αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και να προκάνουμε. Δεν μας διευκόλυνε αυτό το έργο, αλλά καλά τα πήγαμε. Ευχαριστώ πολύ. Good. Well, thank you. Μάλιστα, σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι αύριο ψηφίζουμε σε αυτό, ναι. Αύριο λοιπόν. Ε, ο κύριος Σμιτ δεν ήταν εδώ. Ξέρω ότι είχατε συμμετάσχει στη συζητήση με την κυρία Γκέπχαντ. Εν πάση προσβλέπουμε σε μια καλή δουλειά αύριο και ο κύριος ε, Κλούτσα είχε συνεργαστεί, είχε έρθει να με δει μάλιστα. Και είχαμε πει ότι δεν θα βάλουμε εμπόδια γιατί εδώ ήταν ένα σχέδιο επί του οποίου δουλεύαμε πολύ καιρό και η Επιτροπή επί της αρχής υποστηρίζει. Και πολύ χαίρομαι λοιπόν που η κυρία Γκέπχατ σημείωσε τόσο καλή πρόοδο. Λοιπόν, επόμενο σημείο είναι το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Κόλιν Λάγκεν για ένα νέο φάκελο νομοθετικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο, στις δημόσιες συμβάσεις. Να καλήσω λοιπόν την κυρία αμέσως ε, σε λίγο την κυρία Κόνιν Λάγκεν για τους ε, σκιώδεις η κυρία Γκέπχαρντ Ε, καλύπτεται για, την, για τον κύριο Ταραμπέλα, όχι. Η κυρία Γούλα είναι εδώ, ο κύριος Κρόιτσμαν είναι εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει απαρτία ε. σκιωδών εισηγητών. Έχουμε και κάποιους συναδέλφους από την Κομισιόν, δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει. Α, δεν είναι εδώ ακόμα, λέει ο πρόεδρος. Ωραία θα περιμένουμε να δούμε αν θα έρθει κάποιος από την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Η κυρία Κόλιν Λάγκεν, αν θέλετε να μας ε, παρουσιάσετε τις συμπεράσματά σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς το ίδιο πρόβλημα είχαμε κυρία Κέπχαρτ, πολύ σφιχτό ε, χρονικό πλαίσιο με λίγες δυνατότητες. Λόγω και της τερκουάς εβδομάδας της περασμένης δεν μπορούσαμε να έχουμε επαφές και συναντήσεις. Μερικές ε, γραπτές ανταλλαγές απόψεων. Μια φορά συναντηθήκαμε με την Κομισιόν και μια φορά με τους κοιόδης ηγητές. Και η επόμενη ε, συνεδρίαση είναι στις 17-11 και στις 3-12 14 Εντεκάτου είναι οι τροπολογίες και στις 16 Δωδεκάτου ε, η συζήτηση, ενώ στις 17 Δωδεκάτου ψηφίζει η Επιτροπή μας. Έτσι έχει το χρονοδιάγραμμα. Περί τίνος πρόκειται εδώ. Στόχος είναι η διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Και πρέπει να σας πω εδώ ότι χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα και έχει πολύ μεγάλο νόημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να θέσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης ε, να ε, εκπονήσει ένα νέο πρότυπο σχετικά με στόχο την εναρμόνιση των διαφόρων εθνικών προτύπων για να ε, υπάρχει συμβατότητα των διαφόρων συστημάτων και να γίνει δυνατή ηλεκτρονική τιμολόγηση για να μπορούν οι συμβαλόμενοι στις δημόσιες συμβάσεις ε, με ε, χαμηλή γραφειοκρατία και χαμηλό κόστος να μπορούν να συναλλάσσονται. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα και έχει σίγουρα νόημα. Εκ πρώτη όψεως, η πρόταση είναι σύντομη, είναι κατανοητή, εκ πρώτης όψεως, γιατί εκ Δευτέρας έχουν ανακύψει διάφορα προβλήματα και λεπτομέρειες να σας πω ποια είναι αυτά, όχι όλα, μερικά, τα σημαντικότερα. Μέχρι τώρα έχω δεχθεί και έχω κάνει τροπολογίες, 33 στον αριθμό. Τις έχουν οι σκιώδεις και θα τις συζητήσουμε την άλλη πέμπτη. Και σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι δεν έχουμε προχωρήσει τον έλεγχο όλων των νομικών ζητημάτων είναι ιδέες, προτάσεις και όχι καταληκτικές απόψεις. Δεν έχουμε βρει ακόμα τον τελικό δρόμο ε, που θα είναι και δεσμευτικό και νομικά ισχυρό. Πριν έρθω λοιπόν στις τροπολογίες μου θέλω να σας ευχαριστήσω όλους ειλικρινά και τους κοιόδης που πραγματικά ήσασταν έτοιμοι και τελευταία στιγμή όταν σας ειδοποιούσαμε να έρθετε στις συνεδριάσεις και στη γραμματεία της ΣΥΜΚΟ που μας έχει βοηθήσει τα μάλα. Πραγματικά απίστευτη ήταν η συμβολή της γραμματείας της Επιτροπής και ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα σημαντικότερα θέματα της έκθεσης. Τι προτείνει. να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μία εντολή ε, για ένα πρότυπο το οποίο δεν γνωρίζουμε. Όταν το διάβασα δεν το πίστευα. Ε, ούτε οι συνάδελφοι, ούτε η νομική υπηρεσία τα βασικά στοιχεία στην πρόταση της οδηγίας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Γι' αυτό και εγώ και ε, σε αντίστοιχα με την οδηγία ε, για το φόρο προστιθέμενης αξίας έκανα κάποιες προτάσεις για να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται και τι συζητούμε. Γιατί αυτή ήταν και η κριτική που δεχόμαστε από τους διαφόρους φορείς και τα σωματεία μας έλεγαν ότι αγοράζουμε γουρούνι στο σακί. Τι είναι αυτά που μας ε, προτείνεται. Δεν ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Δεν θέλω να σας πω ότι είναι το απάβγασμα της σοφίας αυτά που ζητάμε, αλλά τα σημαντικότερα. Ε, ένα δεύτερο επίσης σημαντικό είναι η πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει ότι μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας θα πρέπει να έχει μεταφερθεί εντός 48 μηνών. Αυτό ακούγεται πολύ μεγάλο διάστημα, 4 έτη, αλλά όταν δημοσιεύεται η οδηγία, άρα και τίθεται σε ισχύ, ε, δεν θα έχουμε ακόμα τις προτάσεις του ΣΕΝ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης, είπαμε. Δεν ξέρουμε τι θα προτείνει ως πρότυπα και τι θα ισχύει. Και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσο θεωρείτε ότι χρειάζεται η ΣΕΝ. Λέει, α, σιγά, μέσα σε ένα χρόνο. Εκείνοι όταν τους ρωτήσαμε μας λένε 30 με 36 μήνες, άρα τρία χρόνια. Και για την πρακτική εφαρμογή και μεταφορά στα κράτη-μέλη παραμένουν 12 μήνες. Το θεωρώ μάλλον αποκλείεται κάτι τέτοιο, να μπορούν εντός ενός έτους ε, ε αρχές των κρατών μελών να τα εφαρμόσουν σε μικρομεσαίε επιχειρήσεις και σε μικρομεσαίε αρχές. Κάτι άλλο στο οποίο διαφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέει η Επιτροπή ότι η ΣΕΝ ε, θα ε, συμβουλευτεί τους ε, κατατόπους οργανισμούς τυποποίησης. Ναι, εντάξει. Αλλά και είναι εμπειρογνώμονες και δεν σημαίνει καθόλου ότι θα είναι όλα έτοιμα και φτηνά και απλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μιλώ για τα πρότυπα ε, και για τις ε, μικρές πόλεις, τους μικρούς δήμους και κοινότητες. Άρα θα πρέπει να δοθεί ένας χρόνος λογικός στα κράτη-μέλη, όχι 12 μήνες, ακόμα και αν έχουν συνεργαστεί δικοί τους εμπειρογνώμονες, θα πρέπει να δούμε να αρχίσει η προθεσμία από τη στιγμή που θα υπάρχουν τα πρότυπα και μετά. Γιατί ενδιαφέρομαι πάντα, σας είπα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες ε, κοινότητες και δήμους. Οι Γάλλοι λένε ότι έχουν πάρα πολύ μικρά χωριά, πολύ μικρές κοινότητε και αποκλείεται εντελώς να έχουν ε, τη δυνατότητα να τα εφαρμόσουν αυτά μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και κάτι άλλο που για μένα είναι επίσης αποφασιστικό, θα πρέπει να δούμε πώς βοηθούμε για την εφαρμογή των προτύπων και το ποιο είναι το κόστος. Ας πούμε, ε, για μένα δεν είναι αυτό πρόγραμμα απασχόλησης για τους διαφόρους ε, εμπειρογνώμονες σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Να μην αρχίσουμε εδώ τώρα να ε, τροφοδοτούμε αυτό τον κλάδο της οικονομίας με ειδικού που πρέπει να προσλαμβάνουν οι αρχές για να τους τρέξουν τα προγράμματα. Λοιπόν, και από νομική και τεχνική πλευράς. Ο χρόνος δεν φτάνει για να συγκεραστεί με τα πρότυπα, θα το δούμε στη συνέχεια. Το έχω ξαναπεί για τις κεντρικές αρχές 18 ε, μήνες και 36 για τις περιφερειακές ε, και τις τοπικές που αναθέτουν ε, αυτές τις συμβάσεις και τα έργα. Επίσης θα πρέπει να γίνεται και μια μετεξέλιξη πάντα των προτύπων για να ακολουθούν την εξέλιξη της τεχνολογίας ε, και το γίγνεσθε εκεί το, της προφορικής. Επίσης, χρειάζονται και υποστήριξη στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των προτύπων με εκπαίδευση και κατάρτιση υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο να είναι και φτηνό και απλό σε σχέση, και απλούστερο με το, ε, όσα ισχύουν σήμερα. Αλλιώ ο κόσμος δεν θα το υιοθετήσει. Έχει δεσμευτεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Και ε, ε, ε πρέπει να είναι υποχρεωτική εφαρμογή για τον αποδέκτη. Ε, είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώς θα τηρήσει αυτό το χρονοδιάγραμμα και πώς θα σκεφτεί την εντολή που θα δώσει στον οργανισμό τυποποίησης. Δεν λέω ότι δεν έχει γίνει καμιά προεργασία, αλλά θα πρέπει ως νομοθέτες να γνωρίζουμε περισσότερα για το χρονικό ορίζοντα. Ευχαριστώ τους και οδησηγητές για την καλή συνεργασία και είμαι βέβαιη ότι Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και θα προχωρήσουμε αντίστοιχα. Και είναι φιλόδοξο και το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω να είμαστε σε θέση να το τηρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you very much. Ευχαριστούμε την κυρία Κόριν Λάγκεν, λέει ο Πρόεδρος, για την πολύ επικοδομητική εργασία αυτή και που συμβουλευτήκατε τους συναδέλφους. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Κρόιτσμαν έχει στήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Κόλλη Λάγκεν. Ήταν πολύ ευχάριστη η συνεργασία μας. Ε, έχει προετοιμάσει πολύ καλά την έκθεσή της. Συμφωνώ με τα περισσότερα. Θέλουμε κοινά πρότυπα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Χρειάζεται οπωσδήποτε αυτό και στο μέλλον θα πρέπει ε, να μπορεί εκείνο που αναλαμβάνει ένα έργο να εκδίδει τα τιμολόγια ηλεκτρονικά. Έτσι εξοικονομεί και κόστος ε, ο ενδιαφερόμενος στις δημόσιες συμβάσεις. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ε, ότι θα πρέπει το συντομότερο μέσα στην οδηγία να συμπεριλαμβάνονται τα πρότυπα και ε, ε, σύμφωνα με την οδηγία για το ΦΠΑ. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει εύκολα να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα. Τα λέει και η συγκήτρια στις αιτιολογικές σκέψεις. Εγώ θέλω να το πάω ακόμα παραπέρα, να είναι και στο διατακτικό σε ένα νομικά δεσμευτικό άρθρο και να ανταποκρίνεται και στις ανάγκε των περιφερειακών και τοπικών αρχών που αναθέτουν δημόσια έργα. Συμφωνώ με το 18 μήνο για τις κεντρικές κυβερνήσεις και 36 μήνες για τις περιφερειακές αρχές και τις τοπικές ε, που αναθέτουν έργα, όλα αυτά μετά τη δημοσίευση των ε, προτύπων. Ε, 30 μήνες για την εκπόνηση των προτύπων, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά λάβουμε υπόψη ότι είναι περιορισμένη σε πολυπλοκότητα, διότι τα νέα πρότυπα ορίζουν ε, τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου. Έξι μήνες δοκιμαστική φάση, ακούγεται δελεαστική, αλλά δεν έχω καταλάβει από την έκθεση τι μορφή θα λάβει αυτό. Πώς θα δοκιμαστεί αυτό. Δηλαδή θα δώσω ένα σωρό λεφτά ε, οι δημόσιες αρχές για να στήσουν ένα νέο σύστημα το οποίο δεν θα είναι καν σίγουρες εάν θα ε, συνεχιστεί μετά την πάροδο του εξαμήνου. Αυτό δεν ήθιστε να γίνεται ε, ε, επίσης ε, δεν γράφουμε κάτι σε μια οδηγία και παραπέμπουμε στι καλένδε μετά ε, τα πρότυπα εφόσον θα τα έχει εκπονήσει ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνονται από την αρχή στην οδηγία. Συμφωνούμε, θα πρέπει να φροντίσουμε να μειωθούν οι προθεσμίε. Θα τα κάνω όλα αυτά σε τροπολογίες, θα τα υποβάλω, αλλά είμαι βέβαιο ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε καλού συμβιβασμού. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank um, σας ευχαριστώ κύριε Ρούλα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, θέλω να ευχαριστήσω πολύ και εγώ την εισηγήτρια. Να πω το εξή μόνο. Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν καλή. Αλλά δεν ήταν επαρκή η υλοποίηση. Και ήταν τεράστια η πίεση και το άγχος. Ε, και αυτό ε, θα πρέπει να το φτιάξουν με τρόπο που να εφαρμόζεται. Και έρχομαι στις προθεσμίες. Τι γίνεται με τις ηλεκτρονικές συμβάσεις και γενικά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Είναι πολύ μικρές οι προθεσμίες γενικώ και συνήθως και δεν μπορούν να τηρηθούν. Οπότε υπάρχει κίνδυνο να καταραίουν και να αναβαγούν. Ήδη από το 2010 λέγαμε ότι το 50% των δημοσίων συμβάσεων έπρεπε να διεκβερώνονται ηλεκτρονικά. Ναι, σιγά μην το πετύχαμε. Ποτέ δεν έγινε αυτό, γιατί δεν ήταν σωστέ οι προθεσμίε, ήταν υπερβολικά μικρέ. Και να έχουμε μια δοκιμαστική φάση όντω, Δεν πρόκειται για νέα στοιχεία, είναι θέμα συμβατικότητας. συμβατικότητας. Δεν μπορώ να το προφέρω αυτό στα γερμανικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Στην πράξη λοιπόν, να δούμε αν είναι συμβατά τα συστήματα, αν υπάρχουν δυσκολίες με τα όσα σήμερα ισχύουν ε, σε σχέση με την διπλανή χώρα, ας πούμε, ε, ασυνοριακά. Και αυτό το εξάμεινο έχει νόημα, γιατί δεν μπαίνουν νέα στοιχεία, απλώς δοκιμάζονται αν είναι συμβατά με τα υπόλοιπα. Και κατά την άποψή μου αυτό το δοκιμάζει μόνο στην πράξη. Έχω και εγώ αντίστοιχε εμπειρίες με τα πρότυπα. Όταν δίνεις μια εντολή για εκπόνηση προτύπων περισσότερο χρόνο από όσο υπολογίζομαι. Θυμάστε με το θόρυβο στα παιχνίδια όπου είχαμε πει εντάξει είναι απλό το θέμα. 30 μήνε χρειάστηκαν για να αποφασίσουν πρότυπα για το θόρυβο από τα παιχνίδια. Δηλαδή η εκπόνηση προτύπων χρειάζεται, είναι κάτι πολύ χρονοφόρο. Μην πιέσουμε πάρα πολύ χρονικά, αλλιώ ε, διακυβεύεται το σύνολο εγχείρημα. Ευχαριστώ. Good, thank you. Perhaps... Ε, Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κάποια σχόλια και από μένα ως σκιώδης εισηγητής και όχι ως πρόεδρος. Συμφωνώ για τη γενική προσέγγιση με αυτά που έλεγε η κυρία Βούλα Υπήρχε πάρα πολλή δραστηριότητα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση μεταξύ των κρατών μελών ήδη και εδώ προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την καθολική υιοθέτηση του μέτρου. Βεβαίως πολλά κράτη-μέλη χρησιμοποιούν υπαρκτά συστήματα και επομένως αυτό η αρχή της διαλειτουργικότητας είναι πάρα πολύ σημαντική μεταξύ των συστημάτων και πρέπει να Είμαστε βέβαιοι ότι όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να ισχύουν σε όλη τη διαδικασία των συμβάσεων, της παραχώρησης συμβάσεων. Διότι απαιτείται διαφορετικό επίπεδο σημασιολογικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της παραχώρησης μιας σύμβασης και κατά τη διάρκεια της τιμολόγησης. Θα πρέπει να το ενθαρρύνουμε λοιπόν αυτό, την τροποποίηση, ώστε τα δεδομένα που εισάγονται στην όλη διαδικασία να είναι αξιόπιστα και αυτό είναι και η αξία του όλου ηλεκτρονικού συστήματος. Τώρα, νομίζω ότι εδώ πραγματικά το μελετήσατε πολύ καλά, αλλά χρειάζεται μια, αν θέλετε, περισσότερη σαφήνεια στην πρόταση. Υπάρχει, υπάρχουν πολύ τεχνικό, τεχνικοί όροι σχετικά με αυτό το πρότυπο σημαζολογικών δεδομένων, ας πούμε. Είναι δύσκολο να βρει κανείς ορισμό διότι είναι λίγο ε, αυταπόδεικτος αν θέλετε ο ορισμός αυτός, αλλά χρειάζεται κάτι ώστε να μας βοηθάει να το καταλάβουμε καλύτερα. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε επίσης ότι το υποστηρικτικό υλικό θα μας χρειαστεί, εγχειρίδια και οδηγοί, ώστε να οι χρήστες να μπορούν να το χρησιμοποιούν το σύστημα καλύτερα. Όλα αυτά θα βοηθούσαν επίσης, <clears throat> τέλος μάλλον, συμφωνώ και με την ιδέα σας για πιλωτικό χρονικό διάστημα εντός της προθεσμίας. Οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα όπως γνωρίζουμε χρειάζεται μία περίοδο ανάπτυξης και θα, θα βοηθούσε να εξασφαλίσουμε ότι το συνολικό χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνει την απαραίτητη περίοδο ανάπτυξης του συστήματος. Κάνοντας αυτό Νομίζω ότι θα βοηθούσαμε τους χρήστες και θα χρησιμοποιήσω εδώ το παράδειγμα του, του εξυγχρονισμού του τελωνιακού κώδικα και μπροστά σε αυτό το αρνητικό παράδειγμα καλό θα ήταν να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να είμαστε βέβαιοι πότε θα είναι έτοιμο προς χρήση το σύστημα. Αντί να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να βρούμε ότι έχουμε ολιστήσει και έχουμε παρεκκλίνει από το χρονοδιάγραμμά μας και αυτό ίσως είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε και με την Κομισιόν. Αυτά από πλευρά μου. Περιμένουμε όμως τις τροπολογίες σας για να δούμε αν έχουμε πρόσθετα θέματα. Η, η κυρία Βάιλα. Ναι, ο δικός μας κοιόδης σήμερα απουσιάζει μεν, αλλά έχω μια παράκληση σε σχέση με τα όσα είπε η συγγήτρια. Πολύ αναλυτικά. Όλα αυτά που είπατε τα καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Δεν έχω διαβάσει βέβαια το κείμενο. Πολύ λογικά μου φάνηκαν και κατανοητά. Αλλά εγώ έχω την εξή εμπειρία, γιατί είμαι παλιά καραβάνα στο Κοινοβούλιο. Διαπιστώνω, πρόεδρε, το λέω και σε εσά, συνεχώ ότι οι προθεσμίες που θέτουμε εμείς δεν τηρούνται. Όχι επειδή είναι πολύ μικρές, αλλά γιατί δεν, πολύ σύντομε, αλλά γιατί δεν το επιθυμούν τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία. Δηλαδή, ε, για ε, τις ε, πληρωμές για την ανάθεση των αμυντικών συμβάσεων ή για τη Γερμανία, τη μεγάλη ισχυρή χώρα με την εισαγωγή της ΕΠΑ. Είμαστε τελευταίοι, τελευταία στιγμή, τελευταίου δύο μήνες βρήκαμε τα λεφτά για να το εφαρμόσουμε. Παρακαλώ να το λάβετε υπόψη. Ε, είμαι κατ' εξαίρεση σύμφωνη σήμερα με τους φιλελευθέρους, άκουσαν, άκουσαν. Εάν από μόνοι μας ε, επιμικίνουμε, παρατείνουμε ακόμα περισσότερο τις προθεσμίες, φοβούμε ότι τα κράτη-μέλη θα χρονοτριβήσουν όπως το συνηθίσουν ακόμα περισσότερο. Και θα περιμένουμε και 10 χρόνια. Το λέω να το σκεφτούμε. Όλα τα άλλα ε, που είπατε τα βρίσκω πάρα πολύ λογικά, αλλά για τις προθεσμίες έχω αυτή την επιφύλαξη. Διότι δεν είμαστε εμείς οι υπερβολικοί και οι αυστηροί, είναι τα κράτη-μέλη που χρονοτριβούν όλο και περισσότερο. Well, ευχαριστώ κυρία Βάιλα. Είμαι βέβαιος ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμφωνείτε με τους ελεύθερους. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά. Συχνά μάλιστα συμβαίνει. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν το είχα αντιληφθεί νωρίτερα. Έχουμε όμως και τον εισηγητή της Εντροπής των Περιφερειών εδώ, την ε, κυρία Σίγκουστον Λάρσον. Στις 7 Σεπτεμβρίου μάλιστα είχε υποβάλει ένα έγγραφο γνωμοδότησης και θα την καλούσα να μας πει και αυτή δύο λόγια επί του θέματος αυτού και ο κύριος Σταν που αν ακούσαμε καλά το όνομά του από την Κομισιόν είναι εδώ υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Σταν που μάλλον θα μιλήσει η ε, κυρία Λάρσον όμως καταρχάς να μας δώσει τις δικές της, ε, τη δική της προσέγγιση είναι καλό που έχουμε την Επιτροπή των Περιφερειών εδώ, διότι τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών είναι οι βασικοί χρήστες, θα είναι οι βασικοί χρήστες του εργαλείου αυτού. Κυρία Λάρσον, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρίνα Σέφτεν Λάρσον από το Βέρμλαντ, είμαι από την Επιτροπή των Περιφερειών. Εκπροσωπώ λοιπόν τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές της ε, Σουηδίας. Εμείς επικροτούμε αυτή την πρόταση, η οποία θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την σύναψη των δημοσίων ε, συμβάσεων. Όμως, θα θέλαμε να κάνουμε δύο προτάσεις. Καταρχάς χρειάζεται επαρκής χρόνος προετοιμασίας πριν να ισχύσει το σύστημα αυτό και δεύτερον πρέπει να διευκολύνουμε την ε, ηλεκτρονική τιμολόγηση με ε, λογικά, λογικές τιμές, με λογικό αντίτιμο. Υπάρχει το θέμα των σημασιολογικών ε, δεδομένων, υπάρχει το θέμα των τεχνικών εξελίξεων. Πρέπει όμως ε, παράλληλα να εξασφαλίσουμε το ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα λάβει χώρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν θέλουμε λοιπόν να περιορίσουμε ε, τα τεχνικά ε, τους τεχνικούς μορφότυπους ε, που αντιστοιχούν στα σημασιολογικά δεδομένα, πρέπει να προσέχουμε και την αύξηση του κόστους. Εμείς έχουμε ένα παράδειγμα, ηλεκτρονική τιμολόγηση στη Σουηδία, η οποία αντισταθμίζει ε, μεν ε, ε, τα διάφορα προβλήματα κόστους, όμως αυξάνει το διοικητικό άχθος. Και αυτό σημαίνει ότι κάποιες επιχειρήσεις προτιμούν τελικά την έντυπη τιμολόγηση, τη συνηθισμένη τιμολόγηση. Οπότε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υποχρεώνεται κανείς να αρνηθεί μια, ένα τιμολόγιο το οποίο δεν συμμορφώνεται με αυτά τα ε, σημασιολογικά δεδομένα ή με ένα συγκεκριμένο μορφότυπο ε, που θα εγκρίνουμε. Ήδη χρησιμοποιούνται υπάρχουν τα πρότυπα του ΣΕΝ ή του ΆΙΖΟ ε, που είναι οργανισμοί που έχουν εισαγάγει προδιαγραφές για τέτοιου είδους τομείς η πληροφορική υποστήριξη πρέπει να χρησιμοποιείται για τα σημασιολογικά αυτά δεδομένα. Η χρήση διεθνών προτύπων ε, καλή είναι βεβαίως και βέβαια πρέπει να εγγράφεται στο πλαίσιο της ε, συμφωνίας ε, της δημόσιας σύμβασης Χρησιμοποιείται και στον ΠΟΕ αυτό το είδος της τιμολόγηση Για, για την Επιτροπή των Περιφερειών η δυνατότητα διασυνοριακού εμπορίου κατά αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξέρετε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις ε, ε, είναι ραγδαίε και πρέπει να μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε και να τις ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις αναθέτουσες αρχές να γνωρίζουν ε, ποιες ε, είναι οι επιλογές που έχουν σε σχέση με τα σημασιολογικά ε, δεδομένα. Χρειάζεται λοιπόν μία διαδικασία ε, πιστοποίησης ε, και μια διαδικασία ε, που θα ακολουθείται από τις, από τις αναθέτουσες αρχές. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν τη σχέση μεταξύ αυτών των σημασιολογικών μοντέλων και των, των τεχνικών εντύπων, εγγράφων που θα γίνονται δεκτά. Και για να μην χάνουμε και χρόνο στο πλαίσιο τη διαδικασία αυτή, πρέπει να υπάρχει και σχέση μεταξύ ε, των τεχνικών ε, εξελίξεων, αλλά και του γεγονότος ότι έχει γίνει έλεγχος στην πράξη των ε, τεχνικών μορφοτύπων που θα χρησιμοποιηθούν. Πρέπει να υπάρξουν πρότυπα που θα εκπονηθούν. Επικροτούμε βέβαια ήδη τις εργασίες που έχουν, τις εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει από το 2007, η δουλειά αυτή έχει δρομολογηθεί στο πλαίσιο του ΣΕΝ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης. Πρέπει να ε, ισχύσουν τα ε, μοντέλα και ε, στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων. Σε μερικές χώρες ήδη χρησιμοποιείται ηλεκτρονική τιμολόγηση. Έχει αποσταλεί, έχουν αποσταλεί και παραδείγματα αυτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ιδιωτικός και δημόσιος τομέας ε, πρέπει να συνεργάζονται προς διευκόλυνση των δημοσίων ε, συμβάσεων. Και πρέπει και στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών ε, δημοσίων συμβάσεων να, μπορείτε, να μπορεί να χρησιμοποιείται ηλεκτρονική τιμολόγηση. Έτερο πολύ σημαντικό θέμα από πολιτικής απόψεως είναι το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής ε, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η Επιτροπή των Περιφερειών ε, φρονεί <laughs> ότι χρειάζεται μια, να προβλεφθεί μια ε, προθεσμία για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και για τις αναθέτουσες αρχές αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικότερα για τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή των προτύπων, μάλλον την εισαγωγή των προτύπων, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία ε, περίοδος 20 μηνών μέχρι την εφαρμογή των συγκεκριμένων σημασιολογικών μοντέλων και πρέπει να ε, καθορίσουμε τι είδους μοντέλα ε, θα χρησιμοποιηθούν. Αυτό δίνει περισσότερες ε, ευκαιρίες ε, σε όσους θα πρέπει να προβούν στην εφαρμογή των προτύπων αυτών ε, και των σημασιολογικών μοντέλων να μπορέσουν να τα εφαρμόσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να εκφράσουμε την άποψη αυτή της Επιτροπής των Περιφερειών για τη δουλειά αυτή. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για την πολύ χρήσιμη τοποθέτησή σας αυτή που δείχνει και την εμπειρογνωμοσύνη και την ανησυχία των μελλοντικών χρηστών του συστήματος όπως έλεγα. Έχουμε ήδη διανύμει την γνωμοδότηση τη δική σας στα μέλη. Δεν ξέρω πότε θα εγκριθεί επισήμως. Πότε προβλέπετε αυτό μαζί με τις απολογίες. Er Στις 28 Νοεμβρίου είμαστε εν μέσω της διαδικασίας. Στι 28 Νοεμβρίου θα είναι η επόμενη ολομέλειά μα. Δεν ξέρω ακριβώ τι τροπολογίε θα έχουν υποβληθεί ω τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει για την ώρα οι απόψει μα νομίζω συγκλίνουν. Ήταν αρκετά η ευρεία η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Πολλέ περιφέρειες εξέφρασαν την άποψή του. Η διαβούλευσή μα ε, ήταν πάρα πολύ επικοδομητική και η διαδικασία μα έχει δρομολογηθεί, όπω σα είπα και προηγουμένω. Σα ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που προσήλθατε και σε μελλοντική ευκαιρία με μεγάλη χαρά να ανταλλάξουμε και πάλι απόψεις. Να ακούσουμε τώρα τον κύριο Στάμπα για να επανέλθουμε στην κυρία Κόλλιν Λάγκεν και να κλείσουμε το ζήτημα. Εσείς σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να σας πω ποιος είμαι γιατί η πρώτη φορά έρχομαι εδώ σε αυτή, με την ειδικότητα. Είμαι επικεφαλής της υπηρεσίας ε, που ασχολείται ακριβώς με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και μάλιστα είναι τιμή για μένα που στην πρώτη ημέρα της νέας μου λειτουργίας έρχομαι εδώ. Ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Κόλλιν Λάγκεν για την ποιότητα της νομοδότησης και τους κοιόδους ε, εισηγητές για τη δουλειά τους. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο για τη μελλοντική μας δουλειά. Πολλά χρήσιμα εθίχθησεν. Θα δώσω και σε λίγο το λόγο στο συνάδελφο που ασχολείται με το πεδίο αυτό εδώ και καιρό και θα μπορέσει να καλύψει πιο συγκεκριμένα. Αλλά θα ήθελα απλώς ε, καταρχάς εγώ να συνοψίσω αν θέλετε το βασικό μήνυμα, το συνολικό μήνυμα σχετικά με τη δουλειά αυτή. Παρότι πρόκειται για αρκετά τεχνικής φύσεως οδηγία, <clears throat> δεν πρέπει να χάσουμε την βασική έννοια τη εσωτερική αγορά, πίσω από όρου όπω ε, διαλειτουργικότητα που είναι δύσκολο να την προφέρει κανεί, λέει ο μιλητή. στην ουσία κρύβονται συνώνυμα για την εσωτερική αγορά. Αυτό προσπαθούμε να τονίσουμε ότι θα είναι μία ενιαία αγορά για τι επιχειρήσει. Αυτό είναι το σημαντικό και δεν θα πρέπει να χάνουμε το στόχο αυτόν. Τον βασικό αυτό στόχο βεβαίω, και θα πρέπει να συζητήσουμε και όλε τι λεπτομέρειε. Από εκεί και πέρα μιλούμε και για εξοικονόμηση και σήμερα με τα μεγέθη στη διάθεσή μα ε, εξοικονόμηση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για τους επιχειρήσει για τι ε, αναθέτουσε με συγχωρείτε όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα είναι στο κέντρο τη ε, μελλοντική μα συζήτηση και άρα και το χρονοδιάγραμμα είναι σημαντικό. Διότι πρέπει να κινηθούμε σύντομα ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την εξοικονόμηση αυτή παρότι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να είναι προσεκτική για να είναι πλήρω λειτουργικό το σύστημα. Και δεν πρέπει να αποκλίνουμε όμως όσο μπορούμε από το χρονοδιάγραμμα. Η τεχνολογία εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Θα μπορούσαμε να έχουμε και ρήτρες σε και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε την σωστή ισορροπία μεταξύ της σωστής λειτουργικότητας και πλήρης λειτουργικότητας του συστήματος και της ε, ταχείας προόδου, θα έλεγα. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Μπάκτος Ντβόρακ, ο οποίος θα μας ε, αναφέρει πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Θα έχουμε και την, αργότερα ενδεχομένω την ευκαιρία, αλλά θα θέλαμε να σημειώσουμε δύο ή τρία στοιχεία τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να συζητηθούν και στο μέλλον και με τα οποία ίσως να αντιμετωπίσουμε μια δυσκολία ήδη στην φάση αυτή. Σας ευχαριστώ. Όπως είπε ο Νικήτα, να αναφερθώ σε δύο ή τρία σημεία τα οποία είδαμε στην γνωμοδότηση και τα οποία θα θέλαμε να σχολιάσουμε. Υπάρχουν αρκετά σημεία που μπορούμε να δεχθούμε, να συμφωνήσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και αρκετά στοιχεία που ανέφερε ήδη η κυρία Κόλεν Λάγκεν στη συνάντηση. Καταρχάς η δοκιμαστική αυτή περίοδος, το οποίο αναφέρθηκε και από τους κοιόδης συγγητές το όλο θέμα της συμβατότητας, της δημιουργίας του προτύπου και της δοκιμαστικής αυτής περίοδου προτού τεθεί σε λειτουργία. Νομίζω ότι σε αυτήν την ε, χρονική φάση η Κομισιόν ε, θα μπορούσε να εκφράσει πράγματι μια ανησυχία σχετικά με το στοιχείο αυτό, γιατί πρέπει να διατηρήσουμε υπόψη τι ακριβώς προτείνουμε, τι ακριβώς εννοούμε εδώ. Εδώ προτείνουμε ένα πρότυπο, ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, την ανάπτυξή του, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει έναν κατάλογο στοιχείων και την σημασία την έννοιά τους. Το όνομα της επιχείρησης, τον αριθμό ΦΠΑ, την ε, διεύθυνση κτλ. Όταν θα είναι διαθέσιμο το πρότυπο, το πρότυπο αυτό θα πρέπει μετά να περάσει σε μια ηλεκτρονική μορφή μέσω χρησιμοποίησης λογισμικού, είτε άμεσα από τον αποστολέα, ή από έναν πάροχο υπηρεσιών ενάντια αμοιβή. <clears throat> Τώρα, η όλη έννοια της ε, δοκιμής ενός προτύπου, που στην επόμενη φάση θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία, είναι λίγο προβληματική. Διερωτώμεθα πώς θα μπορούσε κανείς να θέσει σε δοκιμασία ένα τέτοιο πρότυπο. Αν είναι σε μορφή λογισμικού να δοκιμαστεί, τότε αν εντομοδίσουμε λάθη, τι είναι, λάθη με το πρότυπο ή λάθη με το λογισμικό το ίδιο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτή την πτυχή. Από την άλλη μεριά, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πολύ μεγάλο τμήμα της δουλειάς θα γίνει επί τη βάση τεχνικών προδιαγραφών που υφίστανται ήδη και σε μεγάλο βαθμό ήδη χρησιμοποιούνται. Επομένως, η ανάπτυξη του προτύπου ή προτύπων χρειάζεται εξακριβώσεις, ελέγχους ε, και δοκιμές. <clears throat> Μας ανεσχεί λοιπόν πώς θα μπορούσε κανείς να το δοκιμάσει αυτό. Αφενός γιατί είναι... Δεν είναι και τόσο απλό, αλλά θα χρειαστεί αφετέρου να έχουμε και μια ηλεκτρονική μορφή που να ε, ε, στη διάθεση των χρηστών. Τώρα για την συμβατότητα με υφιστάμενα συστήματα ή εθνικά πρότυπα, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, κάτι που πρέπει να απογραμμίσει κανεί πιστεύω είναι ότι το πρότυπο που προτείνουμε προς ανάπτυξη δεν είναι καθεαυτό ένα πρότυπο που θα μπορούσε να διαλειτουργήσει με άλλα εθνικά πρότυπα, αλλά θα βοηθούσε στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων, όχι μεταξύ των προτύπων. Θα είναι λοιπόν ένα εργαλείο από τη βάση του οποίου οι χρήστες θα μπορούσαν να αναπτύξουν λογισμικά που θα εξασφάλιζαν τη διαλειτουργικότητα. Δηλαδή δεν θα είναι αυτό το ίδιο που θα εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα, αλλά είναι ένας οδηγός, κάποιες κατευθύνσεις, ώστε να μπορούν τα συστήματα να ευθυγραμμιστούν, αν θέλετε, και να λειτουργούν σωστά το ένα με το άλλο. Ε, πρέπει να είμαστε λοιπόν σίγουροι τι εννοούμε. Τώρα, για το στοιχείο, το κατάλογο των στοιχείων τη εκτελεστική πράξη και κάτι που ίσως νομίζω αναφέρθηκε και στο σχέδιο γνωμοδότηση και από την Επιτροπή των Περιφερειών. Για τον κατάλογο αυτόν είναι κάτι που είμαστε έτοιμοι να το εξετάσουμε ε, ε, στον βαθμό που διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα και την εξοικονόμηση. Είναι κάτι που μπορούμε να το εξετάσουμε λοιπόν. Τώρα, σχετικά με τις εκτελεστικές πράξεις για την αναθεώρηση του προτύπου ή και του καταλόγου ή και της υιοθέτηση του προτύπου, εδώ θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τη διαδικασία προβλέπει ο κανονισμός τυποποίησης, ο οποίος λέει αυτή τη στιγμή ότι το πρότυπο έτσι όπως το έχει αναπτύξει ένας από τους οργανισμούς του τυποποίησης είναι σύμφωνα με τα όσα λέγονται στην επίσημη εφημερίδα και έχουν δημοσιευτεί. Αυτό προσπαθούμε να τηρήσουμε. Προσπαθούμε να το έχουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και αυτή είναι η προσέγγιση που έχουμε προσπαθήσει να αναλάβουμε στην προτινόμενη οδηγία για να προς αποφυγή περί Τώρα, αναγνωρίζουμε την επιθυμία και την ανάγκη του συνομοθέτη να συμμετάσχει στην όλη διαδικασία και μπορούμε να εξετάσουμε πώς θα μπορούσαμε να το εξασφαλίσουμε αυτό σε μελλοντικές συζητήσεις. Ίσως δηλαδή, ε, αν δεν κανεί ε, τον κανονισμό στο άρθρο 11, τον κανονισμό του υποποίησης, όπως ανέφερε και ένας από τους προηγούμενους ομιλητές, αναφέρεται στην πιθανότητα επίσημης αντίρρησης επί προτύπου και αυτό ίσως θα μπορούσε να αναφερθεί. Αισθανόμαστε όμως ε, ότι η προσθήκη των, των εκτελεστικών πράξεων ε, εισάγει μια διαδικασία που προσφέρεται, διατίθεται από τον κανονισμό και με την οποία δεν συμφωνούμε απολύτως και ίσως ε, προσθέτει ένα επίπεδο καθυστέρησης το οποίο με οδηγεί στο τελευταίο που θα ήθελα να θίξω, ακριβώς το χρονοδιάγραμμα. Όπως ήδη ανεφέρθη, Μία από τις βασικές ανησυχίες όπως ανέφερε και ο Νικήτα, ο συνάδελφος, είναι η εξή. Εδώ μιλούμε για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την αναθέτουσα αρχή που θα πρέπει να το χρησιμοποιεί όσο πιο εύκολα και φθηνά γίνεται για να υπερβαίνονται τα όποια εμπόδια ώστε να τιμολογείται μια υπηρεσία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός της ιστορικής αγοράς. Είναι κάτι δηλαδή προς το οποίο θέλουμε να εξασφαλίσουμε ταχύτατη εφαρμογή στο μέτρο δυνατού. Σημειώνουμε βεβαίως ότι δεν μπορεί να υπάρχουν εγγύησει σχετικά με το πότε τελικά θα είναι διαθέσιμο το πρότυπο. Και στο σύνολο της όλης διαδικασίας διαβούλευσης με τους συναδέλφους που είναι υπεύθυνοι για την τυποποίηση κτλ. Μας είπαν ότι το πρότυπο θα μπορεί να είναι διαθέσιμο αρκετά σύντομα και αυτό αναφέρθηκε Επί τη βάση αυτή προτείναμε τους 48 μήνες που θεωρήσαμε ότι επιτρέπουν ένα χρονοδιάγραμμα δύο ετών για την προετοιμασία του προτύπου και άλλα δύο για την εφαρμογή, για την υλοποίηση. Βεβαίως δεν έχουμε εγγύησεις. Γιατί πρόκειται για μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία η ανάπτυξη των προτύπων που ενέχονται πολλοί οργανισμοί και φορείς. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε ευέλικτοι στην διασυνδεσιμότητα ε, τη διαδικασία αυτή ε, με την ανάπτυξη του προτύπου. Αυτό είναι κάτι επί του οποίου μπορούμε να είμαστε ευελικτοί, αλλά το να διαρρέσουμε το χρονικό πλαίσιο μεταξύ κεντρικών, αν θέλετε, αρχών και μη κεντρικών αρχών, δεν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο. Στη διαβούλευσή μας αντιληφθήκαμε ότι η υλοποίηση της ηλεκτρονικής ε, τιμολόγηση ε, είναι τόσο δύσκολη όσο η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού δικτύου. Μπορεί κανείς να εχει διαφορετικέ απόψει, απόψεις, αλλά από κράτη-μέλη μας είπαν ότι η τιμολόγηση προχώρησε ε, το σύστημα το σχετικό, το ηλεκτρονικό, ακόμα και τόσο γρήγορα όσο ένα εξάμεινο. Επομένως εξαρτάται από τις εξελίξει αυτέ και δεν βλέπουμε την ανάγκη να διαρρευθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα μεταξύ κεντρικών αρμοδίων αρχών και μη κεντρικών. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει γρήγορα και εύκολα ενδεχομένω. Υπάρχουν συστήματα διαθέσιμα στην αγορά και η ερώτηση είναι αν κανείς αναπτύξει ένα σύστημα από το μηδέν αυτό είναι η καλύτερη χρησιμοποίηση των πόρων και του χρόνου που έχει στη διάθεσή του. Επομένως θα πρέπει να είμαστε όσο πιο δυνατόν σύντομοι και να αποφύγουμε την περιπλοκότητα. Θεωρούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες να το επιτύχουμε αυτό. Αυτά θα είχα να σας πω προς τον παρόν, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Καλώ ήρθατε για πρώτη φορά εδώ, κύριε Στάμπα. Ελπίζω να έρθετε πολλές φορές, ε, όχι μόνο για αυτή την πρόταση, αλλά και για άλλε που αφορούν τι δημόσιε συμβάσεις. Κυρία Κόλλιν Λάγκ, μήπως θέλει να συνοψίσει και να μας ε, επιβεβαιώσει το χρονοδιάγραμμα. Ναι, θέλω ίσως να διευκρινίσω μερικά σημεία, γιατί μάλλον υπάρχει και παρεξήγηση. Κοιτάξτε, τι λέει η οδηγία. Από τη δημοσίευση αρχίζουν να τρέχουν 48 μήνες. Και πώς θα γίνει αυτό, σε τι ε, αναλύεται αυτό. Μα είπε η Κομισιόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποίηση θέλει 12 μήνε. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, ελέγχεται. Και τα κράτη-μέλη στη συνέχεια έχουν 36. Μέχρι εδώ καλά και είπαμε ότι είναι πολύ ωραίο αυτό το διάστημα. Και μα λέει η ΣΕΝ ποιους 12 μήνε, 30 με 36 θέλουμε. Δηλαδή αν βάλουμε απόλυτε προθεσμίε και μετά χρειαστούν περισσότερο χρόνο για τα πρότυπα, τότε είναι μικρότερο ο χρόνο που έχουν τα κράτη-μέλη στη διάθεσή Γι' αυτό είπαμε να έχουμε ένα ελάχιστο περιθώριο για τα κράτη-μέλη. Εάν μπορεί η Επιτροπή, η ΣΕΝ, και εγώ είμαι πρόθυμη για κάθε συμβιβασμό, ε, αυτή τη στιγμή ε, καταθέσει τα πρότυπα και εγκριθούν, τότε να αρχίσει να τρέχει η προθεσμία που θελήσαμε σύντομη. Ε, ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να εκταθεί πέραν του 48 μήνου. Ναι, να γίνουν όλα γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά και όχι εις βάρος των τελευταίων που είναι η ΟΤΑ, ή οι ε, μικρές δηλαδή αναθέτουσες αρχές ή η μικρή αναδοχή του έργου μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό έχει σχέση με το εξή. Επιτρέψτε μου να πω. Δεν ήξερε και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θέλει να κάνει με την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ε, κατά πώς θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική και τι μορφή θα λάβει ή αυτό που θα είναι ε, κάτι ε, μεταβατικό και ε, από κάποια στιγμή και μετά να μην μπορεί ο παραλήπτης να αρνείται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Μπορεί κάποιοι να έχουν ένα σύστημα εθνικό, ξέρω εγώ, και με εμπειρογνώμονες, παράλληλα οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης σας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην τα συζητούν μεταξύ τους οι τεχνικοί χωρίς καμία συνεννόηση με εκείνους που θα κληθούν να εφαρμόσουν το σύστημα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο αν γίνει. Ξέρω ε, τι λέω, πριν από 16 χρόνια ήμουν δήμαρχος σε μια πόλη ε, και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει ορισμένα τεχνικά να έρχεσαι να τα εφαρμόσει στην πράξη. Χρειάζεται προσοχή εδώ για να μπορέσουμε να έχουμε έλεγχο του συστήματος. Ε, με ενδιαφέρον άκουσα και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφοριών και διάβασα την προσωρινή γνωμοδότηση που δεν έχει εγκριθεί ακόμα, όπως ακούσαμε θα εγκριθεί στις 28 11 θα παρακαλούσα εγκαίρως να μου τη στείλετε για να συμπεριλάβουμε και στη δική μας έκθεση της σκέψης γιατί μέχρι τις 16-12 θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα και θα παραμείνουμε σε επαφή. Για μένα έχει το εξή σημασία, το έχω εξηγήσει και στους Κιώδης, να το πω και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστό και καλό να γίνει αυτό το βήμα, αλλά και οι τελικοί αποδέκτες να το έχουν με διαφάνεια ε, και να μην είναι κάτι υπερβολικά ε, χρονοβόρο ούτε κόστοβόρο, να μην τα επομίζονται όλα οι τελικοί χρήστες, δηλαδή και να μην ε, έχουμε προβληματικές προθεσμίες έτσι ώστε να μπορούσαν να τηρηθούν. Είχαμε και πολύ λίγο χρόνο για την εκπόνηση της έκθεσης. Υπήρξαν και κάποιες νομικές ανομαλίες. Ε, δεν το αρνούμε. Ε, θα πρέπει να τα δούμε αυτά, πώς θα τα διορθώσουμε από νομικής απόψεως και το θεωρώ εφικτό. Γιατί συνήθως όταν αναγνωρίζεις και μόνο ένα πρόβλημα, έχει κάνει το πρώτο βήμα για τη λύση του. Ευχαριστώ. Συνήθω λέω στι περισσότερε περιπτώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κόλιν Λάγκεν. Οπότε, μέχρι τις 14 Νοεμβρίου θα έχουμε την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. 16 Δεκεμβρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες, συμβιβαστικές τροπολογίες. Και στις 17 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε. Βέβαια, ελπίζω να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα αυτό και η Επιτροπή μας. Ελπίζω το Συμβούλιο να σημειώσει πρόοδο επί των θεμάτων αυτών επίσης ε, και ελπίζω να έχουμε συζητήσεις ε, ε, πολύτιμες με το Συμβούλιο ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μέχρι το Φεβρουάριο να δρομολογήσουμε τις, την πρόταση αυτή το συντομότερο δυνατόν. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι η κυρία Κόρι Λάγκεν και η κυρία Λάρσον ε, ε, έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στην ε, διαχείριση των θεμάτων αυτών. Τις ευχαριστώ και τις δύο. Να πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξής μας που αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την ενιαία αγορά αυτών. Έχω το προνόμιο να είμαι εγώ συντάκτης γνωμοδότησης. Ο κύριος Κοφεράτη είναι εδώ, αντιπρόεδρός μας. Ας προεδρεύσω όμως εγώ λίγο ακόμη. Ήρθαν εδώ και οι συνάδελφοι να συμμετέχουν στη συζήτηση, γιατί είναι βασικοί συνάδελφοι αυτοί που μόλις ήρθαν για την ε, πρόταση αυτή. Να τους αφήσω να βγάλουν το παλτό τους. Να βγάλουν λοιπόν τα παλιτά τους ε, οι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκή Επιτροπής. Η κυρία Μπάστο είναι εδώ. Ο κύριος Κρόιτσμαν είναι εδώ. Η κυρία Βερνιό δεν είναι εδώ όμως. Κυρία Γκέπχαρτ. Κυρία Γκέπχαρτ. Evelyn. Evelyn. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Um, uh, Η κυρία Βερνιό δεν είναι εδώ. Μήπως την αντικαθιστά κανείς. Όχι, γνέφει η κυρία Γκέμπχαρτ. Όποιος θέλει να σχολιάσει πάντως, φαντάζομαι θα το κάνει. Θα ήθελα μερικά γενικά σχόλια να κάνω σήμερα. Κατόπιν ε, συζήτησης ναι. με τους κοιόδους συζητητές. Ναι, περιμένω. Λοιπόν, είχα μια πρώτη συνάντηση με τους κοιόδους συζητητές και τους εκπροσώπους τους. Η ομάδα που δουλεύει μαζί μας είναι η κυρία Χάρτιν εδώ, η κυρία Κόλλη εδώ, ο Σεμπάστιαν είναι πάρα πολύ καλή ομάδα μας ε, και πολύ ισχυρή γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο να φέρουμε εις πέρα στη δουλειά αυτά. Μέχρι τις 7 Νοεμβρίου πρέπει να συντάξω τη γνωμοδότησή μου. Επειδή είμαστε επιτροπή υπεύθυνη για τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η δουλειά μας που είναι η οδηγία για τις, ε, οικουμενικές υπηρεσίες, για τις καθολικές υπηρεσίες ε, και τα δικαιώματα των καταναλωτών, πρέπει να καταλάβετε τη σχέση μεταξύ ε, της συγκεκριμένης πρότασης κανονισμού και του τι υπάρχει ήδη στην οδηγία. Και θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί ε, πρέπει να πω ότι εγώ δεν έχω πιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει υπόψη οτιδήποτε ε, είχε αναφέρει ότι θα συμπεριλάβει στην ε, πρότασή της και νομίζω ότι η δικιά μας λεπτομερής ανάλυση, την οποία βέβαια κάποια στιγμή θα μοιραστούμε με την Επιτροπή, είναι μια σημαντική διαδικασία. Πριν όμως μπω λεπτομέρειες. Ε, θα ήθελα καταρχάς να σας ενημερώσω για το γεγονός ότι τώρα έχουμε μια συμφωνία με την, για τη μεθοδιολογία εργασίας ε, σε σχέση με την ε, αρμόδια καθήλυνη επιτροπή, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει, μας έχει στείλει στοιχεία ε, που αφορούν τα δικαιώματα των χρηστών και τις μεταρρυθμίσεις σχετικά με τον τομέα αυτό, όπως επίσης και τις αλλαγές που επηρεάζουν τις άλλες τρεις ε, οδηγίες, αδειοδότηση, πλαίσιο αδειοδότησης ε, και πρόσβασης, που είναι βέβαια αρμοδιότητα της Επιτροπής Βιομηχανίας. Οπότε η πρόταση μου ε, προ την Επιτροπή Βιομηχανία ε, ήταν να αναλάβουμε πλήρη την ευθύνη για όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί είναι στοιχεία για τα οποία είχαμε την ευθύνη αυτή εξ αρχή. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τη δουλειά για όλα αυτά. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που αφορούν, για παράδειγμα, ε, που αφορούν τα δίκτυα και ο Κλάους λένε θα μας πει ορισμένα πράγματα πιο ε, συγκεκριμένα. Αν θυμάμαι μόνο μία πρόταση, μία συγκεκριμένη ρήτρα ε, είναι προβληματική, αλλά η κυρία Ντελκαστήγιο και εγώ θα συνεργαστούμε επί του σημείου αυτού, γιατί νομίζω ότι είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ε, για όλους εσάς. Δεν ήθελα εγώ να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, οπότε θα προσπαθήσω να αναφερθώ κυρίως σε κάποια γενικά σημεία ε, αρχής που νομίζω ότι βρίσκουν σύμφωνους και τους σκιώδεις εισηγητές ε, και μπορούν να το επιβεβαιώσουν άλλωστε και σήμερα εδώ δημοσίως. Φαντάζομαι ότι δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη. Εν όψη ολόκληρου του θέματος ε, και των δραστηριοτήτων της, Ευρωπαϊ... της Επιτροπής μας αυτής για τα δικαιώματα των χρηστών, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πλήρους εναρμόνισης μιας ολόκληρης πτυχής των δικαιωμάτων των χρηστών για τις ε, ε, ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν είναι κάτι το οποίο εγώ ε, το βρίσκω ιδιαίτερα ευνοϊκό. Δηλαδή, θυμάστε ότι είχαμε μια ολόκληρη συζήτηση από πλευράς χρηστών των δικαιωμάτων, ε, δικαιωμάτων των χρηστών. θυμάστε ότι οι οργανώσεις προστασίας καταναλωτών δεν είχαν δεχθεί αρχικά την πρόταση αυτή και ειδικότερα προς τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπου οι καταναλωτές πάρα πολύ εύκολα μπορούν να βρεθούν σε μειονεκτική θέση ε, λόγω καινοτομιών. Η ακαμψία που παρουσιάζει ένα πολύ δεσμευτικό κανονιστικό ε, πλαίσιο προτάσεων από κεντρική νομοθεσία δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι υπέρ ε, των καταναλωτών μακροπρόθεσμα. Μπορεί να υπάρχουν κάποια πλέον εκτήματα βεβαίω στο να, υπάρχει, να υπάρχουν απόλυτα συνεπείς όροι και πιστεύω ότι το 2009 ε, με τις σχετικές προτάσεις δημιουργήσαμε αυτό το πλαίσιο. Είναι όμως σημαντικό, δεδομένου ότι έχουμε ένα ε, σώμα εθνικών ρυθμιστών εντός της δικής τους αγοράς ο καθένας ε, ενεργεί ε, με τρόπο δικό του, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν αυτά τα, στοιχήματα, ή τα συστήματα, οι εθνικοί ε, ρυθμιστικοί φορείς να μπορούν να πάνε πέρα από αυτές τις διατάξεις που αναφέρονται στους στον πυρήνα των κανονιστικών διατάξεων και ελπίζω ότι όλοι θα συμφωνήσετε αν αυτό είναι αντικείμενο τροπολογιών εκ μέρους μου γιατί νομίζω ότι πάντοτε αυτή ήταν η δική μας θέση ε, ως Επιτροπής. Ένα δευτερεύον σχόλιο, το οποίο έχει άμεση σχέση με αυτό, είναι ότι αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε ένα δίκτυο ανεξάρτητων ρυθμιστών ε, που βρίσκονται κοντά στην αγορά και ολόκληρη προστασία συντονισμού των ανεξάρτητων ρυθμιστών με καλύτερο τρόπο ήταν μια πρόταση την οποία η Επιτροπή μας υποστήριξε πάρα πολύ στο πακέτο του 2009 και δεν βλέπω κανένα λόγο να ε, ε παρεκκλίνουμε αυτού, ε, σε αυτό το στάδιο. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής μου φαίνεται ότι το κάνει αυτό όμως και γι' αυτό ε, βρισκόμαστε ακόμα σε ένα εξελικτικό στάδιο. Είναι όμως σαφές ότι οι ρυθμιστές συνεργάζονται πολύ στενά μεταξύ τους, ανταλλάσσουν απόψεις και κατά τη γνώμη μου, επί αυτού του σημείου λεπτομερή πρότυπα ή εναρμόνιση πράγματι μπορεί να λάβει χώρα αποτελεσματικά. Επίσης, ε, δεν συμφωνώ καθόλου με το να δώσουμε με ε, εκτελεστικές πράξεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να ορίσει τις λεπτομέρειες της όλης διαδικασίας. Γι' αυτό έχουμε ε, την Μπέρεκ. Άλλωστε, νομίζω λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές θα είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με αυτόν, λόγω αυτού του, του κεντρικού μηχανισμού. Οι συνάδελφοι που δούλεψαν επί των, ε, της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών ε, θα θυμούνται ότι πέντε χρόνια πριν ε, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό, με την πρόταση αυτή, κυρία Γκέπχαρτ το θυμάται αυτό πολύ έντονα, και θέλαμε να εξετάσαμε την την ε, μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί ήθελε πλήρως εναρμοσμένα δικαιώματα. Ε, όταν εξετάσαμε τότε την αξιολόγηση αντικτύπου, δεν βρήκαμε κανένα αποδεικτικό στοιχείο ε, και μέχρι τώρα σε καμία αξιολόγηση αντικτύπου δεν έχω δει υποστήριξη υπέρ της ανάπτυξης ενιαίας αγοράς ένα, ένα, ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να έχουμε πλήρη εφαρμογή, αυστηρή εφαρμογή όλων των ε, στοιχείων που θα οδηγήσουν σε μια ενιαία αγορά. Και νομίζω ότι κάποιες από τις προτάσεις του κανονισμού αυτού είναι πάρα πολύ λεπτομερείς. Ε, είναι μια μακρο, μικροδιαχείριση τέλος πάντων διάφορων στοιχείων ε, που είναι υπερβολικά λεπτόμερη στις, αρχικές, ε, στις αρχικές μας ε, προτάσεις το 2009 είχαμε συμπεριλάβει πολλά στοιχεία τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τότε είχαμε πρωτοστατήσει γιατί υπήρχαν τότε θέματα για παράδειγμα όπως ε, ε, συγκεκριμένοι όροι συμβάσεων ε, τα οποία δεν τα είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βλέπω ότι τώρα αυτό έχει διορθωθεί στην τρέχουσα πρόταση. Συμφωνεί πλέον με την άποψή μας αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω όμως να εξασφαλίσω ότι η φάση της εφαρμογής είναι απολύτως σημαντική και έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν υπονοεί ότι δεν έχει εφαρμόσει πλήρω κάθε χώρα με αποτελεσματικό τρόπο τι αρχικέ προτάσει που κάναμε το 2009. Όμω, κατά την άποψή μου, δεν ε, νομίζω ότι το είπαν αυτό αρκετά ε, και δεν είναι λόγο αυτό επαρκή για να περάσουμε τώρα σε ε, ε κανονιστικέ ρυθμίσει. Ένα ακόμη θέμα που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά δύσκολο και έχει να κάνει με το πεδίο εφαρμογή τη συγκεκριμένη πρόταση. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση ότι φαίνεται να υπονοεί, αν κατάλαβα καλά από τη διατύπωση τη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι υπάρχουν πολλές λεπτομερείς προτάσεις που αφορούν τους καταναλωτές που θα έπρεπε να ισχύουν για όλες τις συμβάσεις. Όλες, ανεξαιρέτως, για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών. Εμένα αυτό δεν μου φαίνεται ότι είναι, είναι σωστή προσέγγιση. Ε, δεν νομίζω ότι έχει αποδειχθεί το γεγονός ότι ε, οποιοδήποτε χρήστες... Ε, ηλεκτρονικών επικοινωνιών ε, ε, χρειάζονται τέτοιου είδους προστασία ε, ή ότι υπάρχει κάποια ανεπάρκεια της αγοράς ε, στο σημείο αυτό. Στην αρχική μας πρόταση, με τη δική σας υποστήριξη και όντως είχαμε κάνει διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλα γιατί δεν ήταν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως είπα αυτό, ήταν δική μας πρόταση που την προωθήσαμε είχαμε πει οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς να εφαρμόζουν τα στοιχεία δικαιωμάτων των καταναλωτών στις μικρές επιχειρήσεις. Αυτή ήταν μια επιλογή που είχαν στη διάθεσή τους. Είχαμε πει ότι αυτή η διατύπωση είχαμε βρει, εν πάση περιπτώσει, τότε. Τώρα, κατά πόσο αυτό εφαρμόζεται σωστά από τους εθνικούς ρυθμιστικές ε, αρχές, ε, έχουμε ένα σχετικό έγγραφο από την ε, Πέρεκ και βεβαίως ευχαρίστως να το μοιραστώ μαζί σας. Οι, μικρο, οι μικρές επιχειρήσεις μπορεί να θέλουν να επωφεληθούν από κάποιες από, από, κάποιες από αυτές τις προτάσεις, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να παρατείνουμε, να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής στο βαθμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θέλω να σας τα πω όλα αυτά, γιατί αν συμφωνήσετε με αυτά που λέω, αυτό θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις τροπολογίες μου. Τον τόνο των τροπολογιών μου, για να σας το πω διαφορετικά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι εγώ θα ήθελα να ε, υποτιμήσω τη σημασία που έχει όλο αυτό το πακέτο για τους καταναλωτές. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να, ε, να, ε, να μας πει ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να υπερασπιστεί τους καταναλωτές, εγώ θα διαφωνήσω. Όχι, είναι καλύτερα να έχουμε επιτόπου νομοθεσία κοντά στην αγορά, να μπορέσει να λύνει τα προβλήματα στα σημεία όπου δημιουργούνται διάφορα ε, προβλήματα ε, είτε πρόκειται για κάποια τεχνολογική δραστηριότητα, είτε για ζητήματα ανταγωνισμού. Αυτά τα ζητήματα είναι αυτά που πρέπει να λύσουμε ε, στο συγκεκριμένο ε, πακέτο, ας πούμε, συγκεκριμένη οδηγία που αφορά την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτές είναι οι βασικές μου αρχές. Και ήθελα να το πω Γιατί αυτό το θέμα, για παράδειγμα, της ουδετερότητας ε, του ε, δικτύου, ξέρετε πολύ καλά ότι ο ορισμός αυτού δεν είναι πάρα πολύ καλός. Την τελευταία φορά είχα ζητήσει από την κυρία Βίλεν να μας ε, ορίσει τι θα πει αυτό και δεν, δεν έγινε τελικά, δεν ακούσαμε τέτοιου είδους ορισμό. Και έχει σημασία ο ορισμός αυτός, γιατί έχει να κάνει με το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι ήδη έχουμε διατάξεις για τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς ε, να ε, διαχειριστούν ε, την διακριτική τις, τις διακρίσεις όσον αφορά τη χρήση ορισμένων φορέων ε, ή τον αποκλεισμό κάποιων φορέων. Ε, κάτι το οποίο βεβαίω ε, συνιστά διακριτική μεταχείριση. Το θέμα είναι ότι εμεί θέλουμε την αλλαγή μέσω αυτή τη οδηγία ή θέλουμε να έχουμε ένα ισχυρό πλαίσιο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες αλλαγές, οποίε από τώρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Έχει σαχαγεί κάποιε νέε έννοιε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα εξειδικευμένων υπηρεσιών, Εντελώ καινούρια έννοια αυτή στο πλαίσιο ενό ε, ε, νομικού εγγράφου και όλα αυτά σας τα λέω για να είμαι βέβαιη ότι συνεννοούμαστε και ότι καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν είμαι καθόλου πεπισμένος ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουν διατυπωθεί ορισμένα πράγματα σε, αυτό το έγγραφο, ειδικότερα ε, όταν μιλάμε για κανονισμό, ε, δεν είμαι καθόλου πεπισμένο ότι αυτή είναι η σωστή ε, προσέγγιση. Ειδικά όταν μιλάμε για μια ραγδαία εξελισσόμενη αγορά, είναι διαφορετικέ, μάλιστα ταχύτητε με τι οποίε εξελίσσεται ο τομέα αυτό, ε, ανάλογα με τον τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν πριν αποφασίσουμε να επιβάλλουμε ένα ζουρλομανδία για το τι πρέπει να κάνουμε ε, στο μέλλον, καλό θα ήταν να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία, να δούμε τη διατύπωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας. Στρέφομαι τώρα προς τους σκιώδεις εισηγητές ε, να με βοηθήσουν να επεξεργαστώ καλύτερα όλα αυτά τα στοιχεία όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Δεν θα πω σε περαιτέρω λεπτομέρειες γιατί ακόμη τις επεξεργαζόμαστε. Έχουμε κάνει όμως πολύ μεγάλη ανάλυση. Έχω ήδη εξηγήσει την ανάλυση αυτή στους κοιότητες εισηγητές. Ε, έχουμε μάλιστα και ένα έγγραφο σε στήλες για να συγκρίνουμε αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποια από τα θέματα τα οποία ε, τα έχουν θέσει σε εμά οι ρυθμιστικοί φορείς και τώρα έχουμε τέτοια στοιχεία ε, και από τους ρυθμιστικούς φορείς αλλά και από άλλους φορείς και θα χαιρόμουν όλος ιδιαίτερος αν οι σκιώδεις συζητητές μπορούσαν να μας ε, πούν κατά πόσο συμφωνούν με τη γενική μου προσέγγιση γύρω από τα θέματα της εναρμόνισης ειδικότερα να δούμε κατά πόσο μπορούμε πράγματι να βελτιώσουμε σοβαρά αυτή την πρόταση και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι θα ήταν καλύτερα νομίζω αν μας είχε δοθεί η δυνατότητα να, τροπο, να υποβάλουμε τροποποιήσεις σε, αυτήν, σε αυτήν την οδηγία, ε, ειδικότερα από την πλευρά των δικαιωμάτων των καταναλωτών, νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματική αυτή η διαδικασία. Το να συμπεριλαμβάνουμε αυτά τα στοιχεία σε έναν κανονισμό δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό τρόπο. Για το θέμα τη περιαγωγή, για παράδειγμα, με την κυρία Ντελκαστήγιο συνεργάστηκα πάρα πολύ στενά για αυτό το θέμα. Γιατί η χρονική στιγμή αυτής της πρότασης δεν νομίζω δηλαδή ότι θα εγκριθεί πριν από την επόμενη χρονιά. Σίγουρα θα μας πάρει ένα χρόνο. Ίσως θα έπρεπε ήδη να κάνουμε αλλαγές στην τρέχουσα νομοθεσία περί γιατί τρέχουσα νομοθεσία ούτω ή άλλως εκπνέει σε ένα χρόνο. Και κάτι τέτοιο βέβαια δεν μειώνει την πίεση όσον αφορά τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση της νομοθεσίας της περιαγωγής. Ήδη όμως έχουμε ένα σύνολο προτάσεων που τις έχουμε υποβάλει και γι' αυτό καλύτερα να επικεντρώσουμε την ενέργειά μας ε, στο να εξασφαλίσουμε ότι οι προτάσεις που έχουμε ήδη υποβάλει μπορούν να εφαρμοστούν σωστά και αν να δούμε κατά τους επόμενους μήνες αν χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία. Γιατί η αγορά της περιαγωγής ε, εξελίσσεται αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα στάδιο εξέλιξης. Υπάρχουν διάφορα πακέτα που προ... προτείνονται από τις διάφορες ε, εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ λοιπόν η δουλειά της κυρίας Δελκαστήγιο. Γιατί την τελευταία φορά είχαμε συζητήσει ειδικότερα ε, τα μηνύματα κειμένου που πρέπει να στέλνονται στους χρήστες ε, σε σχέση με την περιαγωγή και θέλω να δω πώς έχει εξελιχθεί αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας και με πολύ ε, χαρά θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Πρώτα με την κυρία Μπάστος, την κυρία Μπάστος, μετά ο κύριος Κρόιτσμαν και δεν ξέρω ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ τα πρώτα ε, που θα ήθελα να σχολιάσω. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Χάρμπορ, και την προσέγγιση που μόλις μας υπογράμμισε. Τον ευχαριστώ που συνεργάστηκε ευθύ εξ αρχής ε, με τους σκιώδεις συζητητές ε, επί του, της νομοθετικής αυτής δέσμης. Την Επιτροπή αυτή είχαμε ήδη σε διάφορες περιπτώσεις την ευκαιρία να δούμε την ανάλυση αντικτύπου της Κομισιόν που είναι ουσιώδης σημασίας και να εκφράσουμε τις αμφιβολίες μας σχετικά με την καταλληλότητα του χρονοδιαγράμματος των μέτρων αυτών που προτείνονται. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η ανάλυση αντικτύπου διεξήχθη ώστε να δικαιολογηθεί το επίγον αυτής της νομοθετικής προτάσεως και της υιοθέτησή της και θα ήθελα να το καταστήσω σαφές ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόταση αυτή έτυχε πολλών κριτικών, ομόφωνων σχεδόν, από διάφορους ενδιαφερομένους, μεγάλους, μικρούς, ε, δημόσιους και ιδιωτικούς και απέναντι σε αυτό το σύνολο κριτικής προς το οποίο συμφωνώ θα ήταν ουτοπία να θεωρήσει κανείς ότι αυτό θα υιοθετηθεί στην πρώτη ανάγνωση και εντός της παρούσας εντολής. Τώρα, παρόλο που η Κομισιόν μας λέει ότι αυτό είναι επίγον, αυτό δεν θα πρέπει να μας αποτρέψει από την ε, εντατική εξέταση και ανάλυση των όσων μας προτείνει η Κομισιόν. Στις 24 και 25 Οκτωβρίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ασχολήθηκε με την ψηφιακή ατζέντα και διευκρίνησε ότι είχε αναλάβει αντίστοιχες θέσεις προς αυτές που μόλις λέω και ότι χρειαζόταν μια ενδελεχέστερη ανάλυση ώστε να εγκριθεί και να υιοθετηθεί την κατάλληλη στιγμή μια τέτοια πρόταση. Επομένως λοιπόν θα συμφωνούσα με τα όσα είπε ο εισηγητής μας αυτό που θα ήθελα επίσης αυτή τη στιγμή να κάνω είναι να τονίσω τα εξή σημαντικά σχετικά με την περιαγωγή, με το roaming. Εκπλήσουμε με την προϋπλοκότητα εδώ. Είχαμε εξηγήσει από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαμε δημοσιεύματα στον τύπο από τι αρχέ του Σεπτεμβρίου και εγώ είχα αποκομίσει την εντύπωση ότι εδώ θα πάμε σε ένα κλείσιμο Τη φάση αυτή τη περιαγωγής, αλλά δεν βλέπω αυτό να προτείνεται. Η μόνη περιαγωγή που θα εξαφανιστει οπω όπως βλέπω, είναι από 1η Ιουλίου 2014 για αυτού που δέχονται τηλεφωνήματα. Δηλαδή ακόμα θα υπάρχει κόστος περιαγωγής. Όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό και θέλετε να αποστείλετε SMS, μήνυμα, ή όταν καλείτε σε αυτές τις περιοχές δεν εισάγονται μέτρα χαμηλότερου κόστους ή τιμής και δεν βοηθάει τους καταναλωτές ούτε υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε τέτοια μέτρα. Κάτι διαβάζουμε σχετικά με ένα μια νότη χρέωση 5 cent αλλά νομίζω ότι οι ενώσει καταναλωτών και οι ίδιοι καταναλωτέ θα είναι απολύτω απογοητευμένοι από όλα αυτά. Η Κομισιόν απλώ αυτό περιορίζεται στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων επί εθελουσία βάση να ευθυγραμμίσουν το κόστος περιαγωγή με το εθνικό κόστος από το 2016. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η πρόταση που θα υποβάλει το Κοινοβούλιο θα είναι πολύ πιο φιλόδοξη σε σχέση με το τέλος της περιαγωγής. Εξ αρχής η, το, η ομάδα του ΕΛΚ ε, υπερασπίστηκε τα επιχειρήματα μιας ανάγκης πρότασης πιο φιλόδοξης. Αν είναι να έχουμε μια ρυθμισμένη και ανταγωνιστική αγορά, χρειάζεται ανταγωνισμός. Και όλοι γνωρίζουμε στην πραγματικότητα ότι η παραγωγή έχει ένα κόστος. Η επιβολή λοιπόν της περιεγωγής μέσω νομοθετικής πράξεως θα έχει μια μετακύληση, αν θέλετε, τις επί των καταναλωτών. Διότι θα επιχειρήσουν οι επιχειρήσεις να το εξισορροπήσουν ε, με έμεσους πλάγιους τρόπους, τιμολογώντας άλλου είδους υπηρεσίες. Αυτό συνολικά σαν προσέγγιση προς την περιεγωγή. Δεύτερον, Διαφωνώ και με τα όσα ελέγχθησαν σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Γιατί εκεί θεωρώ ότι η πρόταση θα μπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητική σε κάποιο βαθμό, διότι υπερασπίζει τους καταναλωτές από κάποιες χρήσεις των επιχειρήσεων, όπως ε, τα μακροπρόθεσμα, οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις Έχουμε και άλλες υπηρεσίες, η, μετα... η δυνατότητα μεταφοράς του αριθμού ενό κινητού τηλεφώνου κτλ. Όλε αυτέ όμω, όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να βελτιωθούν και να ευθυγραμμιστούν κυρίω με τα υφιστάμενα πρότυπα επί αποζημίωση και εξασφάλιση τη ε, προστασία των καταναλωτών. Θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητη μία απόλυτη εναρμόνιση υπό την έννοια των βελτίστων πρακτικών και της ε, καινοτομίας. Θα πρέπει να ακολουθούμε πράγματι μια βασική γενική αρχή, αλλά να επιτρέπουμε και ένα περιθώριο ευελιξίας που θα μπορεί να εισάγεται, να εισαγάγεται, με συγχωρείτε, σε εθνικό επίπεδο. Και νομίζω ότι αυτή θα έπρεπε και είναι ε, η προσέγγιση του Ευρωπαίου νομοθέτη. Τώρα, μικρότερη ουδετερότητα. Αν θέλετε, είναι από τις μεγαλύτερες απουσίες, από τα μεγαλύτερα κενά στην πρόταση αυτή. Πρέπει να θυμόμαστε πάνω από όλα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο σε διάφορες περιπτώσεις έχει υιοθετήσει σαφέστατη θέση λέγοντας ότι δεν χρειαζόμαστε συγκεκριμένη νομοθεσία επί της ουδετερότητας του δικτύου Η Κομισιόν ε, είχε βγάλει μια ανακοίνωση θεωρώντας ότι πρέπει να νομοθετήσει στην ε, περιοχή αυτή και πέρυσι ακατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καλύτερο μέσο θα ήταν μια μη δεσμευτική σύσταση. Εμείς το ΕΛΚ θεωρεί ότι η φυστάμενη νομοθεσία πράγματι είναι επαρκή ώστε να εξασφαλίσει την ε, αποτροπή των ε, αποκλήσεων και των παραβιάσεων σχετικά με την ουδετερότητα του δικτύου. Τώρα η Κομισιόν όμως έχει αγνοήσει την επαναλαμβανόμενη αυτή θέση του Κοινοβουλίου και τις προτάσεις που προσπαθούν να εξασφαλίσουν την προάσπιση της αρχής της του δικτύου στο πλαίσιο της νομοθεσίας. Αυτή ε, συνολικά η έλλειψη σημαίνει ότι καταγράφονται, υφίστανται τόσε πολλές καταχρήσει που η χρήση την οποία προσπαθούμε να υπηρετήσουμε έχει θρεβλωθεί. Δηλαδή οι εξαιρέσει γίνονται ταχύτατα κανόνες. Μέχρι στιγμή η έλλειψη πρόσβασης στο διαδίκτυο είχε αντίκτυπο στη διαχείριση ε, του φόρτου μερικές φορές όπως προέκυπτε και από δικατικιστικές αποφάσεις ε, επί της παιδικής πορνογραφίας για παράδειγμα. Και η διασφάλιση της ουδετερότητας του δικτύου είναι... Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που θα μπορούσε να δώσει κανείς. Και υπήρχε μια αρκετά ε, επιθετική λογική πίσω από όλα αυτά, αλλά με την πρόταση αυτή αυτό που καθίσταται σαφές πλέον είναι ότι οι πάροχοι θα πρέπει να αναπτύξουν τις σχέσεις τους με τον καταναλωτή επί τη βάση των δεδομένων που παρέχονται και της προσβάσεως στο δίκτυο. Αλλά αυτό που φαίνεται ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι η εξαίρεση θα μπορούσε, όπως έλεγα, να γίνει ο κανόνας. Δηλαδή, ένας παράοχος να τιμολογεί ειδικέ υπηρεσίες, ειδικέ υπηρεσίες εντός εισαγωγικών, οι οποίες δεν ορίζονται, και ο δημόσιος χαρακτήρας του διαδικτύου θα μπορούσε να απειληθεί. Θα ήθελα λοιπόν Πρόεδρε να συνοψίσω λέγοντας ότι μπορείτε να υπολογίσετε στην πλήρη στήριξή μου ως ε, σκιώδους εισηγήτριας σχετικά με την ε, συνέχιση μιας ε, σαφούς και αντικειμενικής και ενδελεχούς ανάλυσης στο πρόβλημα αυτό. και πρέπει σε κάθε περίπτωση να απορασπιζόμαστε τα δικαιώματα των καταναλωτών και την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς τηλεπικοινωνίας στην Ευρώπη. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάστος. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέγω ευθύ εξ αρχής ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται πάρα πολύ αργά, απελπιστικά αργά και θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν έχουμε αρκετό χρόνο για να ασχοληθούμε επί της ουσίας και με την ισχύα μας με το κείμενο. Βασίζεται μεν στο ισχύο πλαίσιο, αλλά επιφέρει και πολύ μεγάλες αλλαγές και μάλιστα σε πολύ διαφορετικά επίπεδα και πεδία. Και έρχομαι στο πρώτο κρίσιμο σημείο ε, και ερώτημα. Έχει νόημα να τα έχουμε όλα στην ίδια δέσμη όταν γνωρίζουμε ότι ενδεχομένως η οριστική απόφαση δεν πρόκειται να ληφθεί εντό παρούση θητεία σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο, αν τι άλλο. Και μήπω θα πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστέ και να εγκρίνουμε αυτά που είναι εφικτά τώρα και τα υπόλοιπα που θα έχει και επιπτώσει και πιο μακροπρόθεσμε να τα αφήσουμε καλύτερα για να το σκεφτούμε. Γνωρίζουμε τις δομές ε, στις τηλεπικοινωνίες πολύ συχνά είναι ολιγοπόλια αλλά και τα ολιγοπόλια ακόμα έχουν ανταγωνισμό και ιδιαίτερα αυτές οι εταιρείε έχουν δει τις μετοχές τους να μειώνονται πάρα πολύ και έχει να κάνει και με την ανταγωνιστικότητά τους διότι τους αγοράζουν διάφοροι καρχαρίες και αρπακτικά της χρηματαγοράς θα πρέπει να προσέξουμε και οι εταιρείε αυτές να έχουν ε, μια ευκαιρία να επενδύουν και να ε, επενδύουν στις νέες τεχνολογίες. Είχα τη χαρά στην Επιτροπή ε, βιομηχανία, να πάω σε μια αποστολή στη Νότια Κορέα και διαπιστώσαμε ότι οι εταιρείε εκεί είναι στην επόμενη γενιά του γρήγορου διαδικτύου και από έχουμε πόρο εμείς στη Γερμανία από όλα αυτά και φαντάζομαι και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και αυτά τα ζητήματα, ότι έτσι έχει η ζωή. Ε, βέβαια δεν είναι όλο άσπρο μαύρο, στην πρόταση υπάρχουν και θετικά και εκτός από τα αρνητικά. Τα επόμενα χρόνια ε, επίκυνται μεγάλες επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες και ε, θα πέφτει λοιπόν και το κέρδος και ο κύκλος εργασιών τους. Προσοχή λοιπόν, γιατί είναι παγκόσμια η υπόθεση του ανταγωνισμού, να μην αποδυναμώσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Για ε, τη ρύθμιση του ε, ραδιοφάσματος, συμφωνώ, είναι καλή η ρύθμιση αυτή, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία που δεν με βρίσκουν σύμφωνο, έχω επιφυλάξει αν μη τι άλλο για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ιδιαίτερα την δετερότητα του δικτύου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, καταρχήν έχει μια θετική και λογική προσέγγιση. Ερωτώ όμως και προβληματίζομαι πώς ορίζεται τελικά η ιδιαιτερότητα του δικτύου. Λέει να μην υπάρχουν διακρίσεις για άλλους παρόχους. Αρκεί αυτός ο ορισμός. Αν αρκεί καλός. Αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ε, μοντέλα Ε, διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα και ε, τρόπος ε, παροχής υπηρεσιών με μεγαλύτερες ταχύτητες, με διαφορετικές προσφορές, μετατοπίσεις. Προσοχή λοιπόν να μην έχουμε διακρίσεις εις βάρος των εταιριών για να υπάρχει και δυνατότητα εφαρμογής των μοντέλων που έχει κάθε εταιρεία. Αυτά προς το παρόν. Ο Μάλκομ Χαμπ ε, είπε ότι στις 7 του μηνός Νοεμβρίου θα καταθέσει ένα σχέδιο γνωμοδότησης και μετά θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Θα συζητήσουμε με βάση το κείμενό του τι γίνεται και τι δεν γίνεται και ε, να είμαστε μεθοδικοί. Αυτό να μας ενδιαφέρει περισσότερο και λιγότερο η ταχύτητα. Συμφωνώ αλλά το χρονοδιάγραμμά μας επηρεάζεται και από την Επιτροπή Βιομηχανίας. 12 με 13 Φεβρουαρίου θέλει να εγκρίνει την έκθεσή τους, οπότε έχουμε χρόνο να συζητήσουμε τη γνωμοδότησή μας και τη γνωμοδότησή μου. Ελπίζω μέχρι την Πέμπτη θα κάνουμε πολύ καλή δουλειά, γιατί έχω μια ισχυρή ομάδα που δουλεύει από αυτού. Αλλά σίγουρα είναι ένα δύσκολο ζήτημα και βασιζόμαστε στην εμπειρογνωμοσύνη σας. Θέλει κανεί άλλος να πάρει το λόγο. Α, συγγνώμη, δεν σας είδα που μπήκατε. Ε. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Ε, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Φερχέν. Ε, θέλω να συμφωνήσω με πολλά από όσα παρετήρησε ο Μάλκομ Χάρμπο. Έχουμε εδώ μια πρόταση που θίγει ένα τομέα πάρα πολύ περίπλοκο και θα έχει και επιπτώσεις και συνέπειες που ενδεχομένως να μην έχουν ακόμα μελετηθεί επαρκώς. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα που προτείνονται εδώ ε, στον κανονισμό δεν ξέρουμε ακριβώς ε, τι τελικές συνέπειες θα έχουν. Το χρονοδιάγραμμα. Νομίζω αναφέρθηκε εκτενώς. Λυπούμε που κατατέθηκε τόσο αργά, ενώ προς το τέλος της θητείας μας η πρόταση αυτή και ε, μας πιέζει αντικειμενικά να λάβουμε μια ταχεία απόφαση για ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά χρειάζεται σοβαρή και σχολαστική μελέτη και για τους ορισμούς. Χρειάζεται να κάνουμε συζήτηση περισσότερη από αυτό το εξάμεινο που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι το τέλος της ε, κοινοβουλευτικής θητείας, εν πάση περιπτώσει και στο Κοινοβούλιο να μας προβληματίσει αυτό. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι συνέχεια και έχουμε ευτυχώς ε, συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει δυνατότητα να συνεχιστεί μια έκθεση. Δεν καταστρέφεται όπως γίνεται στα Εθνικά Κοινοβούλια, δεν καταραίει η έκθεση επειδή αλλάζει το Κοινοβούλιο, Αναλαμβάνει ο ίδιος ή άλλος ηγητής και ε, προχωρεί η προσπάθεια. Ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε ήταν ακριβώς η ουδετερότητα του δικτύου και ιδιαίτερη ποιότητα των υπηρεσιών και πραγματικά εδώ οι επιπτώσεις ενδεχομένως πώς να να ε, μην έχουν μελετηθεί επαρκώς, ακριβώς επειδή είναι κανονισμός ας πούμε αυτός που προτείνεται. Δεν έχετε καταλάβει μάλλον ε, τι συνέπειες θα έχει. Μόλις έρχομαι από το φόρουμ διακυβέρνησης του διαδικτύου ε, που πρόσφατα συζητήθηκε για αυτό το θέμα των περιορισμών στο διαδίκτυο και πώς επηρεάζει αυτός τις υπηρεσίες, γιατί στην Ευρώπη και για αυτά τα θέματα είμαστε φάρος, υπόδειγμα για άλλες περιφέρειες του κόσμου που έχουν στραμμένο το βλέμμα τους επάνω και δεν θέλουν να υπάρχουν διαφορές, προτεραιότητες περιεχομένου στο διαδίκτυο, ταξινόμηση, κατηγορίες. Γιατί πραγματικά ε, αληθορίζουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες περιφέρειες ε, του κόσμου και άλλες υπηροί και έχουν επικρίνει πολύ στη συζήτηση την πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακριβώς για την ουδετερότητα που δεν ορίζεται ακριβώς και επαρκώς, αλλά και άλλες γραφές που κάνετε για τη μη διάκριση να μην υπάρχει δυνατότητα tailoring, blocking και άλλες τέτοιες υπηρεσίες ε, που αυτό το αξιολογούν θετικά. Αλλά οι specialized services τι είναι, ειδικέ υπηρεσίες, ξεχωριστές ιδιαίτερες προσφορές σε ένα νέο τοπίο μηντιακό με προσφορές όλο και περισσότερο όχι τόσο ε, οριζόντιας ε, ολοκλήρωσης αλλά κάθετης. Δηλαδή κάποιος που παρέχει τις τηλεπικοινωνίες παρέχει και περιεχόμενο και πρόσβαση στο δίκτυο και έτσι συνδέονται ορισμένα πράγματα που μέχρι τώρα ήταν ε, ε, αποσυνδεδεμένα και υπάρχει υπερσυγκέντρωση ε, της δραστηριότητας σε μια εταιρεία, πράγμα που σημαίνει και ολιγοπόλιο και περιορισμό του ανταγωνισμού και στο περιεχόμενο και σε κάποιες άλλες μορφές του διαδικτύου. Νομίζω ότι είναι έκθεση ετσεβερίας για το επιγραμμικό εμπόριο και τις ε, παραγγελίες για τη μη διάκριση στο διαδίκτυο για να μπορεί ο κάθε έμπορος να προσφέρει τα προϊόντα του στο δίκτυο και να μην κάνει προεπιλογή ο πάροχος του δικτύου ή ο πάροχος ε, της υπηρεσίας αυτής. Θέλει προσοχή η μη διάκριση, η ε, ελεύθερη αγορά, η δίκαιη αγορά θα πρέπει να είναι δεδομένη και στο επιγραμμικό εμπόριο. Γιατί σε ορισμένε θέσει και αρκετέ θέσει του κειμένου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωράνε βελτιώσει. Και θα ήθελα να ακούσω και τι άλλε επιτροπέ που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Ξέρω ότι η Επιτροπή Πολιτισμού είναι και αυτή ε, έτσι, δυσαρεστημένη από το χρονοδιάγραμμα και μάλιστα ακούστηκε και εντονότατη κριτική σχετικά. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Κάποιο άλλο θα ήθελε το λόγο. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιο θα ήθελε να σχολιάσει από του δύο στα όσα ακούσαμε ήδη. Ρομπέρτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. πραγματικά χαιρόμαστε που η Επιτροπή αυτή εξετάζει πολύ σοβαρά το όλο ζήτημα. Βεβαίως και σημειώνουμε την κριτική σας, δεν μας εκπλήσει, είναι και μέρος των, της δουλειά σας, των καθηγόντων σας. Και παρότι δεν έχουμε δει τη δουλειά που έχετε κάνει, είναι προφανές ότι είναι μια ενδελεχής εξέταση που θα βοηθήσει την αρχική μας πρόταση, την αρχή μας δουλειά. Επίσης ε, ε, μας ικανοποιούν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Όχι μόνο διότι το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η δέσμη αυτή χρειάζεται εντατική εξέταση προς έγκαιρη έγκριση, υιοθέτηση, αλλά και υπό την έννοια των καταναλωτών των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Κινείται δηλαδή το Συμβούλιο σε μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση, αν θέλετε, γιατί λέει στην παράγραφο 5 ότι η αντιμετώπιση του κατακαιρματισμού, η αποτελεσματικός ανταγωνισμός και οι ιδιωτικές επενδύσεις μέσω ενός προβλέψιμου και σταθερού νομοθετικού πλαισίου είναι κρίσιμη σημασία, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη ένα ποσοστό ευελιξίας ώστε να αναλάβουν περαιτέρω μέτρα προστασίας του καταναλωτή. Από τα συμπεράσματα αυτού του συμβουλίου που παρέθεσα προκύπτει ότι και η Κομισιόν πρέπει να το λάβει υπόψη τη, καθότι το Συμβούλιο χαιρετίζει ένα κοινό, την ανάγκη ενός κοινού νομοθετικού πλαισίου σταθερού, αλλά με κάποιο βαθμό πρόσθετης εθνικής προστασίας. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το στοιχείο ή στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, εμείς το λαμβάνουμε υπόψη μας και η Επιτροπή σας σίγουρα είμαι βέβαιος θα το λάβει υπόψη της. Ε, τώρα, ο βαθμός του κατακαιρματισμού που βλέπουμε στην Ευρώπη είναι πραγματικά ανησυχητικός. Εγώ τα τελευταία χρόνια μετακινούμε μεταξύ των χωρών και οι ιστορίες φρίκης που ακούω είναι πολλές που μου έχουν μεταφερθεί και που έχω δει για πολύ υψηλού λογαριασμούς ανευπροειδοποίησης, ε, περίεργες και μυστικές ε, και καθόλου προφανείς ε, συνθήκες, ε, ε, ε, διατάξεις της συμβάσης, αλλά η πραγματικότητα της υλοποίησης εις το πεδίο είναι πάρα πολύ διαφοροποιημένη. Μπορεί να επικρίνεται την μέγιστη εναρμόνιση προς την οποία στοχεύομαι και από ό,τι φαίνεται από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ούτε το Συμβούλιο δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο αλλά αυτό που έχουμε προβλέψει στην πρότασή μας, θα μπορούσε κανείς να το δει και ως τυποποιημένο τρόπο κατά τον οποίο θα έπρεπε να μεταχειριζόμαστε τους καταναλωτές στην, στην Ευρώπη, διότι οι αποκλήσεις που βλέπουμε δεν είναι αποδεκτές. Σε μερικά κράτη-μέλη προστατεύονται οι καταναλωτές επαρκώς και σε άλλα καθόλου. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Και θα ήταν και ανησυχητικό αν η προστασία των καταναλωτών πήγαινε σε κάποια ακραία επίπεδα, που να που τελικά να ήταν τροχοπέδι για την πρόσβαση στην αγορά των επιχειρήσεων το οποίο θα εμείωνε τελικώς την ανταγωνιστικότητα και τελικά και τις επιλογές που θα είχαμε για τον καταναλωτή λέει ο μιλητής. Επομένως η ομοιόμορφη προστασία είναι σημαντική, η μέγιστη εναρμόνιση είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε βεβαίως. Για την ε, ουδετερότητα του δικτύου. Είναι περίπλοκη η συζήτηση. Στην πραγματικότητα όμως το 36% των καταναλωτών στην Ευρώπη ε, υποφέρουν από αυτό το, τη διακοπή ε, και την παρεμπόδιση των, των προσφορών που τους διατίθενται. Ε, το πλαίσιο δεν προχωρεί όσο θα έπρεπε ώστε να δίνει τις ε, δυνατότητες στον νομοθέτη να επιβάλλει διατάξεις που να αποκλείουν αυτό το throttling που γίνεται την παρεμπόδιση σε αυτές τις προσφορές που θα έπρεπε να έχουν οι καταναλωτές. Από την άλλη πρέπει να αναγνωρίζουμε και τις εθνικές συνθήκες και για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες αφήνουμε στους, στις ρυθμιστικές αρχές σε ποιο βαθμό θα επιτρέψουν οι ειδικευμένες υπηρεσίες, διότι αυτό είναι ένα απόσπαστο και αναπόφευκτο κομμάτι της συζήτησης της, ε, και της προεπιλοκότητας συζήτησης ε, για την ουδετερότητα του δικτύου, συζητείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις κάτω χώρες, που είναι από τις λίγες χώρες που έχουν υιοθετήσει τέτοιου ότι οι ρυθμιστικές αρχές του κράτους μέλους θα πρέπει να έχουν την εξοδότηση να αποφασίζουν ποια είναι η χρηστή ισορροπία στις εξειδικευμένες υπηρεσίες, το οποίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι των, ε, του διαδικτύου, όπως έλεγα, για των υπηρεσιών. Τώρα, επαναλαμβάνω, Πρόεδρε, ότι ευχαριστούμε πολύ για τις παρατηρήσεις σας, εκτιμούμε το ε, έργο που κάνετε και θα προσβλέπουμε σε οποιοδήποτε άλλο ε, σχόλιο, πρόταση, σύσταση και περιμένουμε να δούμε και το σχέδιο γνωμοδότησής σας. Με ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι κινούμαστε προς μία βιώσιμη λύση. Όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα μη συνεπούς εφαρμογής των δικαιωμάτων των καταναλωτών και δεν νομίζω ότι κανείς θεωρεί ότι το να αλλάξουμε τη λέξη από σε κανονισμό αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε επιτόπου. Ε, μπορούμε πολύ περισσότερα να κάνουμε γιατί έχουμε ήδη ρυθμιστές ε, που συνεργάζονται ε, σε ένα κοινό μοντέλο, κάτι το οποίο το έχουμε λιγότερο στα δικαιώματα των καταναλωτών που είναι πολύ περισσότερο κατακαιρματισμένα τα πράγματα και την παραπλανητική διαφήμιση και πολλούς άλλους τομείς που θα μπορούσα να παριθμίσω. Εκεί που διαφωνώ με εσάς και την ομάδα σας είναι ότι έχουμε ήδη ένα καλό πλαίσιο το οποίο ε, δημιουργήσαμε το 2009 μαζί. Και το γεγονός ότι υπήρχε κακή εφαρμογή δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αλλάξουμε σε κανονισμό το πλαίσιο αυτό, γιατί αυτή δεν είναι η σωστή λύση κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να σκεφτούμε πού είναι οι αδυναμίες του συστήματος, ε, μπορούμε να αναθεωρήσουμε κάποιες ε, απαιτήσει που υπάρχουν στις οδηγίες, αλλά καλύτερα να συνεργαστούμε για να είναι καλύτερη η εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Γι' αυτό προτείνω στην Επιτροπή ε, στην Επιτροπή μου να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, να μην πάμε από οδηγία σε κανονισμό, γιατί ουσιαστικά μεταφέρεται έτσι η ευθύνη από τους ανθρώπους ε, που πρέπει να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά ε, για τους χρήστες που είναι οι ίδιοι ρυθμιστές. Εκεί είναι η βασική μας διαφορά και πιστεύω ότι οι καταναλωτές ε, μάλλον συμφωνούν, θα συμφωνούσαν περισσότερο μαζί μας όσον αφορά την κωδικοποιημένη ορολογία που χρησιμοποιείται ε, στην πρόταση. Ελπίζω να έχουμε λοιπόν μια καλή πρόταση, ε, σωστή, η οποία θα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα των καταναλωτών, ε, τα περίπλοκα θέματα, τα πιο δύσκολα σημεία που θεωρείται ότι είναι τα πιο ε, σοβαρά και πρέπει να λυθούν. Ούτως ή άλλως προφανώς θα μας ξανάρθετε για την επόμενή μας ναι. συζήτηση. Πολλή δουλειά έχουμε που αρχίζει αμέσως μετά το τέλος της ε, συνεδρίασης της σημερινής. Θα δουλέψουμε όσο αργά σήμερα για να συμπεριλάβουμε όλα τα στοιχεία. Στις 7 Νοεμβρίου θα υποβάλω την έκθεσή μου για μετάφραση. 27 ε, ε, Νοεμβρίου θα έχουμε μια ακρόαση για το θέμα αυτό. Θα εξετάσουμε τη γνωμοδότησή μου στις 28 3 Δεκεμβρίου προθεσμία τροπολογιών, 9 ε, εξέταση τροπολογιών, συμβαστικές 12 και ε, τον Ιανουάριο στη συνεδρίασή μας θα εγκρίνουμε τη δική μας γνωμοδότηση και ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι μέχρι το Φεβρουάριο, τότε που η Επιτροπή Βιομηχανίας θέλει να ψηφίσει τη δική της, ε, γνωμοδο... τη δική της έκθεση. Το θέμα της ουδετερότητας των δικτύων είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το δουλέψουμε γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία στην οδηγία δικαιωμάτων των χρηστών ε, που έχουν να κάνουν για παράδειγμα περισσότερο με ε, στοιχεία της οδηγίας πλαισίου. Έχουν να κάνουν με αυτά περισσότερο τα θέματα και υπάρχουν και κάποιες διατάξεις για την ε, ε, χονδρική πρόσβαση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα που αφορούν ε, τα, ε, τις συμβάσεις που δεν αφορούν τόσο τα θέματα των δικαιωμάτων των κριστών, αφορούν κυρίως τις συμβάσεις αυτές καθεαυτές μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα. Ένα ακόμη θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Ο Τζουζέπε Μεμόντι είναι εδώ και η ομάδα του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τους καλωσορίζω. Είναι εδώ ο εισηγητής μας, ο Ανδρέας Φάμπ. Ποιοι άλλοι σκιώδες είναι εδώ, για να δω. Αντικαθεστά κανείς ε, τον κύριο ε, Γκαρσία Χαμόν. Οι Σοσιαλδημοκράτε λάμπουν δια τη απουσία του σήμερα το απόγευμα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τέλο πάντων, συγγνώμη που το λέω αυτό δημοσίω, απλώ είναι μια παρατήρησή μου. Ο κύριο Σφαμπ και εγώ λοιπόν, εμά είμαστε μόνο. Γιατί και εγώ είμαι σκιώδη συζητητή για το θέμα αυτό. Ε, να δώσω λοιπόν στον Ανδρέα το, το λόγο για να μα παρουσιάσει, ε, παρουσιάσει την άποψή του για τι ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους στο σχέδιο εκτισής μου. Ειλικρινά, μεγάλο ευχαριστώ. Πολύ καλές προτάσεις, χρήσιμες και που βελτιώνουν το κείμενο. Ταυτόχρονα όμως διαπιστώνω ότι υπάρχει ευρύτατη συμφωνία και συνένεση για την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει το σχέδιο έκθεσης. Βέβαια, ως πολιτικός μπαίνει κανείς στον πειρασμό όταν ακούει τέτοιες ιστορίες σαν το σκάνδαλο της NSA ε, να αναστατώνει τον τύπο ε, προσπαθεί να συνδέσει ο κάθε πολιτικό το θέμα του και με αυτό. Ε, αλλά στην Επιτροπή μας τουλάχιστον ε, έτσι, για μακροπρόθεσμους ε, σκοπούς ε, δεν έχουμε μπει σε τέτοιους πειρασμούς, έχουμε αντισταθεί αρκετά. Οπότε καλό θα ήταν να παραμείνουμε στο στόχο μας και στη μακροπρόθεσμη θεώρηση. Και Βέβαια μπορεί να συνδεθεί και με τα πρόσφατα και τα επίκαιρα γεγονότα. Αυτό που μας ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει όσο γίνεται πιο ανθεκτική και να έχει όσο γίνεται μεγαλύτερη αντίσταση ε, εναντί ε, κάθε είδους ε, επιθέσεων, επιδρομών και ιδιαίτερα οι λεγόμενες κρίσιμες υποδομές. Αυτό το δείχνουν και οι πολλές τροπολογίες της έκθεσής μου. Αυτό που μας ενδιαφέρει τελικά είναι ε, το πεδίο εφαρμογή. Έτσι, πού βρίσκει εφαρμογή αυτή η οδηγία. Είναι πάνω από 200 τροπολογίες μου. Πρόκειται για κάποιους παρόχους υπηρεσιών που θέλουμε μου προκειται για καποιου παροχους υπηρεσιων που θελουμε εμεις να τους επιφορτήσουμε με το καθήκον να τηρούν ε, κάποια πλαίσια. Και ε, θα πρέπει να υπάρχει και ένας λόγος ρυθμιστικός. Γιατί. Και ο λόγος ποιος είναι είναι ε, πολύ ευαίσθητε οι υποδομές ή κρισμότητα τέτοια, όπως λέμε τώρα σε μοντέρνα γερμανικά και ξέρουμε ότι είναι η κρισιμότητα τέτοια ε, ώστε ε, κινδυνεύουν οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν ο νομοθέτης θέλει να παρέμβει και πρέπει να παρέμβει. Γι' αυτό από την αρχή ήδη στο σχέδιο εκθεσής μου επικεντρώθηκα πάρα πολύ σε αυτή την έννοια της κρισιμότητας της οδηγίας. Υπάρχει αυτή η έννοια ε, στην Ευρώπη ήδη και αναφέρω τις κρίσιμες υποδομές ε, και οπωσδήποτε και στην παρούσα οδηγία. Τώρα, στο πεδίο εφαρμογή, βέβαια, είναι ανοιχτά πολλά ερωτηματικά. Τι γίνεται με την κοινωνία της πληροφορίας τη λεγόμενη. Εγώ πρότεινα να επικεντρωθούμε στις κρίσιμες υποδομές μόνο, το είπα και προηγουμένως, και τι γίνεται με τους παρόχους υλικού και λογισμικού, ε, hardware και software, διότι δεν είναι καθόλου εύκολο όταν έχεις ένα ευαίσθητο κρίσιμο ε, σύνολο υποδομών. Είναι δύσκολο να ε, προμηθεύεσαι κάθε φορά ε, το υποχρεωτικό ε, υλικό και λογισμικό που σου υπαγορεύει η οδηγία. Για την αστική ευθύνη, αυτό που προτείνει ο κύριος Γκαρσές Ραμόν, σκιώδης ηγητής ε, των σοσιαλιστών και δημοκρατών, αλλά και η κυρία Έγκστρομ, προτείνουν κάποια πράγματα που για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί κινδυνεύουμε να κάψουμε μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Ε, δεσμεύουμε και βάζουμε διάφορες υποχρεώσεις σε όλους τους κατασκευαστές ενώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι εκείνοι που χειρίζονται τις κρίσιμες υποδομές. Νομίζω ότι λίγο το παρακάνουμε εδώ. Επίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τελικά δεν θα έχουν ε, εναλλακτικές προτάσεις ε, στην προμήθειά του στην αγορά λογισμικού και υλικού. Δεν μπορούμε να τους δέσουμε τόσο πολύ τα χέρια και ε, ενδεχομένω για τις μικρομεσαίες να χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα. Άλλο στοιχείο του πεδίου εφαρμογή θα βάλουμε και τη δημόσια διοίκηση εδώ. Βεβαίω στα κράτη-μέλη υπάρχει τεράστια ποικιλομορφία της ένταξης κρισίμων υποδομών στο πεδίο εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Δεν είναι πάντα αυτό γεγονός. Κατά την άποψή μου η δημόσια διοίκηση, με τη στενή έννοια, το στενό κράτος, γιατί περί αυτού πρόκειται, καταρχήν δεσμεύεται, ακριβώς επειδή είναι δημόσια διοίκηση, δεσμεύεται λέγω να ε, τηρεί ε, αυτές τις απαιτήσει για τις κρίσιμες υποδομές. Αλλά Εάν θέλετε οπωσδήποτε να υπενθυμίσουμε στις δημόσιες αρχές ότι είναι καθήκον τους, δεν με πειράζει, αρκεί να μην το θεωρήσουν σκόπελο στο Συμβούλιο τελικώς. Και αν στόχος μας είναι η οδηγία αυτή να εγκριθεί, αν γίνεται, ε, κατά τη διάρκεια της θητείας, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και αυτά τα στοιχεία και τη στάση μας απέναντι στο Συμβούλιο. Αλλά δεν πειράζει, μπορούμε να το βάλουμε ως πολιτικό αίτημα. Επίσης, το επίπεδο της κρισιμότητας νομίζω θα πρέπει να το ε, αποφασίζουν τα κράτη-μέλη, να επιτρέπεται και έτσι θα επιτρέπονται και διάφορα στάδια επέμβασης. Αλλά να υπάρχει ένα ε, ενιαίο πρότυπο βασικό και από εκεί και πέρα το κανονίζουν τα κράτη-μέλη. Το επόμενο, να πούμε ότι για τις τηλεπικοινωνίες υπάρχει ήδη υποχρέωση ε, υποβολής κάποιων στοιχείων και δηλώσεων. Γι' αυτό δεν εμπίπτει στην παρούσα οδηγία. Ο κύριος Γκαρσές Ραμόν το βλέπει κάπως διαφορετικά από τους Σοσιαλιστέ και δημοκράτες, αλλά ε, για μας δεν καταργούνται ε, καθόλου με την παρούσα οδηγία κάποιες υποχρεώσεις αναφοράς από κάποιους κλάδους. Το αντίθετο θέλουμε εμείς. Υπάρχει κάποια στοιχειώδης ε, εναρμόνιση, ας πούμε, έτσι ώστε να ξέρουν οι εταιρείε ε, πώς να προσανατολίζονται και τι διατηρείται και τι καταργείται, που δεν καταργείται. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πώς συνδυάζεται η παρούσα οδηγία με την οδηγία που υπάρχει για την προστασία των δεδομένων ή με τον κανονισμό. Αυτή η οδηγία λοιπόν και η οδηγία προστασίας δεδομένων και ο βασικός κανονισμός θα πρέπει να βαθίζουν χέρι-χέρι και οπωσδήποτε να αποφύγουμε επικαλύψεις αλλά και ελλείψεις. Γι' αυτό δεν θέλησα σε καμία περίπτωση να αναμειχθώ ε, στο πεδίο του βασικού κανονισμού και νομίζω και η κυρία Έγκστρομ το θέλει αυτό. Είναι σωστή η προστασία των δεδομένων, αλλά υπάρχει ξεχωριστή ε, οδηγία και κανονισμός και δεν είναι του παρόντος δεν έχει καμία σχέση η παρούσα οδηγία με την προστασία των δεδομένων. Αυτό που μας ενδιαφέρει μόνο είναι να εξασφαλιστούν, επαναλαμβάνω, οι κρίσιμες υποδομές. που μπορεί αυτό να αφορά και κάποια προσωπικά δεδομένα, αλλά σε πρώτο λόγο και κύριο αυτά ρυθμίζονται αλλού. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα εδώ είναι οι κρίσιμες υποδομές. Αλλά, αγαπητοί συνάδελφοι, η οδηγία αυτή δεν θα πρέπει να μπει στο ψυγείο εκεί που υπάρχουν ήδη κάποιες ρυθμίσεις σε κάποια κράτη-μέλη από το 1995 η οδηγία ε, για την ιδιωτική ζωή ε, στο διαδίκτυο. Μπορούμε όλα αυτά να τα συνδυάσουμε και να τα χωρίσουμε όμως για να ξέρουμε ξεχωριστά τι ισχύει στο βαθμό που υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση ή ε, που επηρεάζει το ένα νομοθέτημα το άλλο, νομίζω είναι ξεκάθαρα. Η ΕΝΙΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονούν ένα εντύπω για να αντιμετωπίζουν από κοινού και με απλό τρόπο ενδεχόμενες ε, κυβερνοεπιθέσεις. Ε, να τις δηλώνουν, εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα, Πρόεδρε, υπάρχει και συνεργασία των κρατών μελών δεν βοηθάει να έχει υπερβολικές εξουσίες ε, επέμβασης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα ζητήματα των κρατών μελών. Αλλά θα πρέπει το Συμβούλιο να καταλάβει ότι θα πρέπει ε, όλοι να καταβάλουμε μια κοινή προσπάθεια για να έχουμε υψηλότερο επίπεδο προστασίας στον κυβερνοχώρο. Και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν και να ανταλλάζουν απόψεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ένα τελευταίο, Πρόεδρε. Έχουν έρθει και πολλές τροπολογίες που υπερβαίνουν το πεδίο της ασφάλειας του δικτύου και της πληροφόρηση για την ασφάλεια. Και αυτό θα παρακαλούσα να το σκεφτούμε αυτό. Είναι συγκεκριμένο το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Τώρα, γιατί να εισαγάγουμε κάποια θέματα που ουσιαστικά δεν έχουν σχέση με το πεδίο αυτό. Τώρα, Πρόεδρε, δεν θα σας εκπλήξει αυτό που μόλις αναφέρατε εσείς, η ιδιαιτερότητα του δικτύου, net ε, ε, ε, neutrality. Αυτό έχει να κάνει με την οδηγία για τις τηλεπικοινωνίες. Δεν έχει καμιά δουλειά εδώ. Και να μην παραφορτώσουμε την πρότασή μας με παράλληλες ρυθμίσεις που το μόνο που θα κάνουν να μας φέρουν σε νέες δυσκολίες. Το άλλο επίσης εύλογο ερώτημα είναι αν θα εισαγάγουμε ένα γενικό καθολικό δικαίωμα για πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες εντάξει, ας πούμε ότι είναι θεμελιώδες δικαίωμα αυτό, αλλά δεν έχει καμία σχέση ε, σε αυτή την οδηγία που ασχολείται, επαναλαμβάνω, με τις κρίσιμες υποδομές και τη δική τους ασφάλεια. Επίσης, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού ή η ένταξη ιδιαίτερα ευάλωτων χρηστών κτλ. Επίσης δεν έχει καμιά δουλειά εδώ, παρόλο που θα το επιθυμούσαν ορισμένοι συντάκτες τροπολογιών. Αποδέκτες της οδηγίας αυτή είναι εκείνοι που χειρίζονται τις κρίσιμες υποδομές. Και τι δουλειά έχουν οι ευάλωτοι χρήστε και οι κοινωνικά αποκλεισμένοι δεν χειρίζονται τέτοια συστήματα. Οπότε ας μην ανησυχούμε. Και ένα τελευταίο είναι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Υπάρχει η διατιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Δεν θα πρέπει να συγχαίουμε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με την πρόληψη ή την αποτροπή του εγκλήματος. Λοιπόν, άλλο πράγμα είναι η δικαιοσύνη που διώκει το έγκλημα, το ηλεκτρονικό και άλλο πράγμα είναι οι δραστηριότητες ορισμένων ξέρω εγώ, μυστικών υπηρεσιών που θα πρέπει να ελέγχονται περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν και θα πρέπει, επαναλαμβάνω, στις δύο περιπτώσεις να έχουμε ξεχωριστές αστικές δομές, αστικές που, και πολιτικές που θα συμμετέχουν και θα συνεργάζονται πέρα από των διοκτικών αρχών ε, για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια στο διαδίκτυο και στον κυβερνοχώρο. Ξέρω ότι θα βρούμε απέναντί μας κάποια κράτη-μέλη. Ε, δεν με νοιάζει, είμαι πρόθυμος να συγκρουστώ ε, μαζί τους και με τις εταιρείες διότι έτσι κι αλλιώς ξέρουν εταιρείε ότι μπορούμε με διάφορες μυστικές υπηρεσίες ε, έχουν πρόσβαση σε αυτές μέσω φιλικών τους υπηρεσιών σε άλλες χώρες κτλ. Γι' αυτό ε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχουμε χωρίσει και οργανωτικά τις πολιτικές δομές πέρα από τις διάφορες ε, υπηρεσίες πληροφοριών, μυστικές υπηρεσίες ή ιδιοκτικές αρχές ενώ ε, για την ποινική αντιμετώπιση, τη, τη δικαστική. Και ένα τελευταίο. Βέβαια έχει ρόλο να διαδραματίσει ο οργανισμός ενίσα, αλλά έχει ένα πεδίο ο δικό του ε, ε, δράσης και δεν μπορούμε, πιστεύω, να δεχθούμε τις τροπολογίες του κυρίου Πουπάκη που ζητούν επέκταση των αρμοδιοτήτων. 19 του μηνό Νοεμβρίου θα το συζητήσουμε και στις 11 Δεκεμβρίου και ελπίζω αρχές Ιανουαρίου, Πρόεδρε, βοηθήστε με με την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ήτρε και ΛΥΜΠΕ. Κανονικά αρχές Ιανουαρίου, λέω, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε για να μπορέσουμε και μαζί με το Συμβούλιο να συμφωνήσουμε κατά τη διάρκεια της παρούσης και περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να μου πούν και οι ηγητές αν έχουν τίποτα παραπάνω από τι τροπολογίε που έχουν καταθέσει και γενικά είμαι αισιόδοξο ότι θα βρεθούμε σε ένα καλό δρόμο και θα επιτύχουμε μια καλή λύση. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, που ηγηθήκατε τη προσπάθεια αυτή τη δύσκολη και τη αφέστατη ε, τοποθέτησή σα σε αυτό το φάκελο. Λοιπόν, έχουμε δύο σκιώδει συζητητέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Αντρέα ε, για την ε, πολύ καλή δουλειά που έκανε. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Ήδη μας παρακολουθεί η NSA. Άρα γιατί να εστιαζόμαστε επί αμερικανικών προτύπων αντί να μην δημιουργούμε ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε ίσως μια μέρα να είμαστε ανεξάρτητοι από όλα αυτά τα αμερικανικά συστήματα και επιχειρήσει, Λέω μήπω. Επίσης έχω ερώτηση. Γιατί αποκλείουμε την δημόσια διοίκηση. Όταν μιλούμε για ζωτική σημασία σε υποδομή και θα έλεγα μάλιστα μεταφοράς ενέργειας κυρίως, Υπάρχει επίσης και το ζήτημα των μικροεπιχειρήσεων και μικροοντοτήτων, οι οποίες θα έπρεπε να αποκλείονται διότι είναι τόσο μικρές που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ζωτική σημασία πληροφορίες ώστε να πρέπει να βαραίνει ακόμα περισσότερο το όλο ζήτημα. Ελπίζω επίσης να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για ένα σύστημα reward ένα σύστημα παροχής κινήτρων αν θέλετε προς τις επιχειρήσεις ώστε να τους, να τους αποδίδεται μια, ένα βραβείο αν θέλετε εφόσον είναι, καταφέρνουν να έχουν λιγότερους ελέγχους να τους παρέχουμε ένα κίνητρο μια επιβράβευση, μια αναγνώριση αν θέλετε, σχετικά με, την, ε, με τον τρόπο που λειτουργούν και για την ασφάλειά τους. Τώρα, οι περισσότερες ε, τροπολογίες που είχα ήταν ευθυγραμμισμένες με την, ε, προς την πρότασή σας και εγώ ελπίζω πραγματικά να βρούμε μια λύση για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον, τον Ιανουάριο. Λέω μιλητής, ευχαριστώ τον ε, κύριο Μάντες κάποια σύντομα σχόλια από πλευράς μου διότι ως σκιώδης είχα υποβάλει κάποια σύντομα σχόλια τροπολογίες σε γενικές γραμμές με ικανοποίηση απολύτως η δουλειά σας νομίζω ότι τις βελτίωσατε ακόμα περισσότερο και εγώ τουλάχιστον ε, άτλησα από την εμπειρία μου επί της οδηγίας ιδιωτικότητας και σχετικά με τις παραβάσεις, ε, σχετικά με την ε, προστασία των δεδομένων για τους καταναλωτές και πώς χειρίζομαστε αυτές. Γιατί πρέπει να είμαστε σαφείς ότι η όλη διάσταση της διαφάνειας είναι σημαντική και γίνεται όλο ένα και πιο σημαντική, αλλά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ίσως να έχουμε πολύ σημαντικά δυνητικά προβλήματα. Κάποιος πρέπει να, είναι, να προσέξει να μην ε, δημιουργήσει σύγχυση η οποία θα μπορούσε να επιδεινώσει τα πράγματα. Επομένως αυτό το ενιαίο σημείο επαφής το οποίο θα μπορούσε να συντονίσει και να διαβιβάσει πληροφορίε σχετικά με την ευαισθησία συγκεκριμένων πληροφοριών ή την συγκεκριμένε παραβιάσεις είναι μια σημαντική πτυχή και άλλη μια πτυχή που θεωρώ ότι είναι σημαντική είναι το πόσο θα είχαν οι βασικοί χρήστες υποδομής την διάθεση να είναι ανοιχτή ο ένας με τον άλλον. σε σχέση με τη διαχείριση εμπιστευτικών στοιχείων, διότι αν είχαμε μία επίθεση, μία συγκεκριμένη παραβίαση, θα έπρεπε να ειδοποιούνται και άλλοι φορείς, αν θέλετε, ώστε να λαμβάνουν ε, μέτρα αμήνης που να συμπληρώνουν το ένα το, άλλο. Και σχετικά με τις ανησυχίες πρώιμης απελευθέρωσης πληροφοριών, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα ζωτικό επίπεδο δραστηριότητα ώστε να μα κάνει να ανησυχεί, να ανησυχούμε, με συγχωρείτε. Αλλά νομίζω ότι όλη η κατεύθυνση είναι ε, ένα πρώτο βήμα, δηλαδή να κάνουμε όλη αυτή την πρόταση πιο ρεαλιστική, αν θέλετε, πιο χρηστική, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα νομοθετικό πλαίσιο και να πάμε όλοι μαζί σε κάποια πρώτα ελάχιστα πρότυπα και, αν, και να δούμε κατά πόσον θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τους πολίτες μας και από αυτού νομίζω ότι έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά. Εάν λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε κάποιες συζητήσεις με τα κράτη-μέλη μετά την ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο, καλώς, Αλλά βέβαιως θα πρέπει να δούμε και ποιες θα είναι οι τάσεις της ελληνικής παιδείας της πρόοδου με το φάκελο αυτό. Αυτά είχα να πω ως ισκιώδης Ξαναβάζω το καπέλο του Προέδρου και ρωτώ, κάποιο άλλο θα ήθελε το λόγο. Ε, κάτι θα θέλατε να προσθέσετε κύριε Μάντες παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι σωστό. Μιλούμε στην Ευρώπη για one-stop shop, ενιαίο ε, σύστημα μάλλον μίας βαθμίδας, ενός βήματος. Αυτό ήταν κάτι που ξέχασα να αναφέρω προηγουμένως και νομίζω ότι είναι σημαντικό. Πάντοτε με χαρά καλωσορίζω τον Τζουζέπε Αμπαμόντε εκπροσωπώντας την Κομισιόν. Δεν ξέρω τι έχει να πει για την έκθεση Σβάμπα. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους τους ε, συναδέλφους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο και να εκφράσω την ικανοποίησή μου με τη γενική κατεύθυνση και το ύφο τη εκθέσεω. Υπάρχει σύγκληση μεταξύ της ε, πρώτης του Ανδρέας και της αρχής πρώτης Κομισιόν και της κυρίας Δεκαστήγιο της Ήτρε. επομένω νομίζω ότι γενικά καλά κινούμαστε. Τώρα η έκθεσή σα, συμπεριλαμβάνει πολύ ενδιαφέρουσε και ορθέ προτάσει και ιδέε σχετικά με την ανάγκη ή τη δυνατότητα των κρατών μελών να ορίζουν άνω της μίας αρχής εθνικός NIS, με συγχωρείτε, και για το ενιαίο σημείο επαφής ώστε να ενθαρρύνεται και να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών προς, όλα αυτά συμφωνούμε. Επίσης ε, συμπεριλαμβάνει κάποιες ε, καινοτόμες και χρήσιμες ιδέες για τις ε, προϋποθέσεις και συνθήκες κοινοποίησης και για την ευθύνη. Και επειδή ο κόσμος τούτος δεν είναι τέλειος, να σας πω ότι υπάρχει και ένα σημαντικό σημείο διαφωνίας μεταξύ μας, ιδιαίτερα επί του πεδίου εφαρμογής και για τη διαχείριση του συστήματος κινδύνου, μάλλον επί του συστήματος διαχείρισης κινδύνου. Συμφωνούμε λοιπόν με την ε, αποκοπή, αν θέλετε, των δημοσίων διοικήσεων και των βασικότερων επιχειρήσεων του διαδικτύου και αν μου επιτρέψετε Πρόεδρε, δύο λεπτά, να πω τα εξή σχετικώς. Όλοι είμαστε υπέρ της αφήνειας δικαίου και της βελτίωσής της, ώστε να διευκρινίσουμε ή να αποσαφηνίσουμε αυτήν την έννοια των internet enablers, των διευκολυντών του διαδικτύου που είναι επιχειρήσεις που διαρματίζουν ρόλο όλο και πιο ζωτικό στα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της κοινωνίας μας. Και ως ελάχιστο θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνουμε στη διαχείριση κινδύνου υποβολή εκθέσεων ή συναγερμού, κρουσμάτων και των σχετικών παρόχων των υπηρεσιών. Την, το περιεχόμενο, μάλλον τις πλατφόρμες ανταλλαγής γνώσεως και περιεχομένου, τους παρόχους ηλεκτρονικού εμπορίου, τους τελικούς χρήστες, των πόρων που είναι απαραίτητοι για την ασφάλεια και την ε, λειτουργία του διαδικτύου, δηλαδή σημεία ανταλλαγή, ε, ονόματα domain, περιεχόμενα κτλ. Συμφωνώ λοιπόν ότι ίσως η έκθεση δεν είναι το πρότυπο της αφήνειας και της καθαρότητας, αλλά ενδεχομένως αυτά θα μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε. Αλλά κάτι ακόμα που είχα αναφέρει, αλλά θα επαναλαμβάνω για πάντα, είναι ότι υπάρχει ένα σημαντικό θέμα εδώ ισορροπίας, ισότητας, ισότιμων κανόνων παιχνιδιού. Είστε ένας από τους πατέρες της μεταρρύθμισης τηλεπικοινωνιών και γνωρίζετε ότι υπό το 30α οι παραδοσιακοί πάροχοι υπόκεινται στις προϋποθέσεις NIS. Επομένως, θα ήταν μια χαμένη ευκαιρία να μην έχουμε τις ίδιες προϋποθέσεις και για τις ε, κυρίαρχες επιχειρήσεις του πεδίου. Και μιλώ για επιχειρήσεις όπως τη Skype ή τη WhatsApp, αν ακούσαμε καλά, που δεν υπόκεινται στις παραδοσιακές διατάξεις του άρθρου 13 και όχι 30α διορθώνει ο Δερμηνέας. Να ολοκληρώσω ε, βεβαιώντα τον κύριο Μάντερς ότι αυτοί οι φορεί που αποκλείονταν στην αρχή τη πρόταση ακόμα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογή. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο για την σαφή απάντηση που μα δώσατε στα σημεία αυτά. Να δώσω το λόγο λοιπόν στον Αντρέα Σουβάπ για να συνοψίσει. Νομίζω ότι έχουμε το χρόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπούμε λίγο που κανεί δεν θέλει να με χαρακτηρίσει εμένα ιδρυτή πατέρα, παρόλο που ακόμα είμαι στο ηλικιακό όριο να έχω παιδιά, τι να κάνουμε. Ε, υποστηρίζω αυτά που είπε ο Τζουζέπε Βαμόντε μόλις. Είναι σαφές ότι πολύ μικρές επιχειρήσεις έτσι και αλλιώς εξαιρούνται και από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως θα πρέπει να επιβραβευτούν οι ίδιοι που το έπραξαν. Ένα αυτό. Δεύτερον, αυτό που είπε ο Τόιν Μάντερς, να επιβραβεύονται εκείνες οι εταιρείε που δεικνύουν σοβαρή συμπεριφορά. Συμφωνώ απολύτως, αλλά αυτό είναι μάλλον εθνική υπόθεση. Είναι θέμα ε, της εθνικής ε, εποπτικής ρυθμιστική αρχής που εκείνοι κάνουν τον έλεγχο. Θα δούμε πώς μπορούμε να τους συμπεριλάβουμε. Συμφωνώ με τη γενική ιδέα πάντως. Όλα αυτά στα αγγλικά. Και επίσης ευχαριστώ πολύ Μάλκομ που εσύ Κοντζάν Πρόεδρος κάθισες μέχρι τέλους της συνεδρίας αυτής. Είσαι και σκιώδης ηγητής. Και ε, χαίρομαι που συμφωνείς με τις κοινέ ε, τροπολογίες συμβαστικές που προτείναμε από κοινού και δεν ε, λες ότι θα πρέπει να βελτιωθεί περισσότερο ακόμα. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε ορισμένες διαφορετικέ αντιστάσεις στα κράτη-μέλη και επανέρχομαι σε αυτό που ρώτησε ο Τόιν ε, Μάντερς. Γιατί εξαιρείται η δημόσια διοίκηση. Το παραδέχτηκα δημοσίως. Πρέπει να γίνει αυτό διότι εν μέρει αυτό ορισμένα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο θα το θεωρούσαν τεράστιο ε, πρόβλημα. Και επίσης εγώ θεωρώ, και έτσι το ερμηνεύω, ότι από τη φύση του το κράτος το ίδιο ε, θα πρέπει να θωρακίζεται απέναντι στις επιθέσεις του διαδικτύου. Δεν λέω ότι να εξαιρούνται. Ξέρω ότι και στην Επιτροπή Βιομηχανίας ε, υπάρχει σφοδρή επιθυμία να συμπεριληφθεί. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Και επίσης στην Επιτροπή Ήτρε ζητούν οι συγμένες εταιρείες ε, κάπου να αναφέρεται αυτό τουλάχιστον σε μια αιτιολογική ε, πρόταση ότι στους ετήσιους ισολογισμούς τους θα πρέπει να αναφέρουν αυτό το στοιχείο της προστασίας από τις επιθέσεις ε, στο χώρο. Αυτά. Μήπως να μας θυμίζατε το χρονοδιάγραμμα ε, της ψηφοφορίας σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία Ελεκτρινά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιρετική συνεργασία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ηγηθήκατε αυτού του θέματος. Ε, χαίρομαι που θα σημειώσουμε πρόοδο. Πρέπει να υπάρξει πρόοδος παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες ανησυχίες ε, από άλλες δραστηριότητες που αφορούν τα θέματα προστασίας δεδομένων, για παράδειγμα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, με τα, ζητήματα ε, που έχουμε μπροστά μας. Μετά τα Χριστούγεννα θα ασχοληθούμε ξανά με αυτό το θέμα, γιατί το Σφάμπ, ο θα ασχοληθεί με τις συμβιβαστικέ τροπολογίες και πρέπει να λάβει τις τροπολογίες Επιτροπής ε, Βιομηχανίας που θα ψηφίσει 16 Δεκεμβρίου και 14 ε, ή 28 και 27 και 28 ε, Νοεμβρίου θα ψηφίσει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Οπότε πρέπει να τα συγκεράσει όλα για τις συμβιβαστικέ τροπολογίες. Εμείς θα ψηφίσουμε το σύνολο του πακέτου και των στοιχείων που θα έχουμε συμπεριλάβει από τις υπόλοιπες ε, ε, επιτροπές. 22 ή 23 Ιανουαρίου θα γίνει αυτό. Αν όλα πάνε καλά λοιπόν, ελπίζω να λάβουμε όλες τις πληροφορίες πριν από τα Χριστούγεννα ε, να πάμε όλοι σε διακοπές και μετά από τα διακοπές των Χριστουγέννων θα είμαστε όλοι πολύ πιο φρέσκοι και θα καταλήξουμε σε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο συμβαστικών τροπολογιών ε, και να τις έχουμε και μάλιστα ως δώρο για το νέο έτος ελπίζω έτσι να πάνε τα πράγματα, αλλά ο Ανδρέας Σουάμπ είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να μας ε, φέρει αυτό το ε, περίπλοκο τελικό προϊόν. Ελπίζω να τα καταφέρνει. Αυτά για σήμερα, τα απόγευμα. Ευχαριστεί ο Πρόεδρος και τους διερμηνείς. Ολοκληρώσαμε τη συνεδρίασή μα σε 5 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα. Αύριο 9 η ώρα το πρωί θα συνεδριάσουμε και πάλι. Θα συζητήσουμε για ε, πρώτα απ' όλα την έκθεση για την ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων του Πάμπλο Αρία Ετσεβερία, τμήμα της δουλειά μας για την ψηφιακή οικονομία. Μετά θα ψηφίσουμε από τις 10 παρατέταρτο μέχρι τις 11 και 4 και έχουμε άλλα δύο θέματα του κυρίου Κοφεράτη. Και το απόγευμα θα αρχίσουμε 3,5 ώρα σας υπενθυμίζω, 3,5 για, με την ακρόαση για τα οργανωμένα ταξίδια. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.